και δεν θα υπάρχει καμία υπέρβαση. Οι διερμηνείς σας πληροφορούν με τα λύπης ότι συνεχίζεται η εργασιακή διαμάχη με τη διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις νέες συνθήκες εργασίας που αποτέλεσε το αντικείμενο προειδοποίησης για περιακή κινητοποίηση. Η ποιότητα της διερμηνίας για τους ευρωβουλευτές και τους Ευρωπαίους πολίτες κινδυνεύει. Δυστυχώς λόγω της εργασιακής διαμάχης η διερμηνία θα σταματήσει ακριβώς όπως προβλέπεται στο πρόγραμμα στις 21 και 45. Δεν έχουμε ε, διερμηνία στα ε, Μαλτέζικα και στα Γκέιλικ. Λοιπόν, έχουμε και ψηφοφορίες που θα είναι σχετικά χρονοβόρες. Σας παρακαλώ να καθίσετε. Λοιπόν, καταρχήν διορισμός των εισηγητών. Η Σιλβίν Βον Κάουφμαν είναι η συγγήτρια για την πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου για θέματα σε σχέση με, ασφάλεια, με την ασφάλεια κατά τους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Η κυρία Κιέγγε από τους σοσιαλιστές είναι συγγήτρια για την πρόταση κανονισμού για τη δημιουργία ε, ενός ευρωπαϊκού δικτύου ε, αναδιατύπωση Σεσίλια Βίκστρεμ από τους φιλελευθέρους. Με συγχωρείτε, είναι, ε, γίνεται λίγη φασαρία. Σας παρακαλώ καθίσετε. Βίκστρομ, φιλελεύθερη, είναι η συγγήτρια ως προς τον κανονισμό για τις, ε, για τις κοινωτικές στατιστικές για τη μετανάστευση. Μαρτίνα Άντερσον η για τις διατάξεις της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Και τώρα, ως προς την ερώτηση προς το Συμβούλιο Οδηγία 2002 κάθετος 19 για την ανθρωπιστική βοήθεια η οποία δεν πρέπει να ποινικοποιηθεί μετά από την απόφαση των συντονιστών στις 24 ε, Μαΐου για την ε, διακίνηση των μεταναστών και την ποινικοποίηση του όλου θεσμικού πλαισίου ε, έχει συμφωνηθεί μία προφορική ερώτηση μεταξύ ομάδων και θα συζητηθεί στην Ολομέλεια του Ιουλίου. Σύμφωνα με, τον, με το άρθρο 128 κάθετος 5. Συμφωνείτε? Εντάξει. Ναι. Ε, δεν δέχομαι να εργαστούμε μόνο στα αγγλικά. Δυνάμει του 158 παράγραφος 1 μπορώ να το ζητήσω και θα το θίξω στη διάσκεψη των Προέδρων. Ευχαριστούμε. Για αυτούς που δεν άκουγαν, πρόκειται για την οδηγία για την πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια. Θα θέλαμε να μας κοινοποιήσετε την άποψή σας. Λοιπόν, πέρα από αυτά, έχουν εγκριθεί οι προτάσεις των συντονιστών ως προς τις ε, κατεξιοδότηση πράξης. Θα ήθελα να με ακούσετε στις Μαΐου η Επιτροπή ε, ε, έλαβε υπόψη συγκεκριμένες, μια συγκεκριμένη οδηγία για τις τεχνικές προδιαγραφές και στις 6 Ιουνίου το Συμβούλιο αποφάσισε να μην αντιταχθεί σε αυτή την κατεξιοδότηση πράξη. Επίσης, δυνάμει του κανονισμού 273 και 111-2011 για, τους, για τις πρόδρομες ουσίες ναρκωτικών υπάρχουν... Ε, με συγχωρείτε για τις ε, πρόδρομες εκρηκτικές ουσίες θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ε, προδιαγραφές με βάση θα πρέπει να λάβουμε αποφάσεις με βάση τα ταξιδιωτικά έγγραφα και η ΛΥΜΠΕ στις 15 Ιουνίου 2018 έλαβε υπόψη αυτά τα δεδομένα. Εάν θέλετε να προβάλλετε αντίθεση, αυτό θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 22 Ιουνίου στις 12. Μπορείτε, σας παρακαλώ, να έχετε και έτοιμες τις κάρτες σας για την ε, ψηφοφορία που επίκειται. Βάιντεν Χόζερ. Έρχεται η κάρτα του. Επί του παρόντος δεν την έχει. Σας παρακαλώ, έχετε τις ε, κάρτες σας. Εάν τις έχετε στην Ολομέλεια κάποιος να μεταβεί, να τις παραλάβει. Λοιπόν, Αυτά ως προς τις κατεξουδότηση πράξεις Έχουμε και ένα άλλο θέμα σε σχέση με τους μετανάστες στη Μεσόγειο. Έχετε το λόγο. Ε, δυστυχώς οι πιο ευάλωτοι πολίτες, οι πραγματικοί πολίτες βρίσκονται σε κίνδυνο. Δεν μιλάμε μόνο για αριθμούς βρίσκονται σε πολύ δυσχερή θέση και μετά από αυτά που ακούσαμε στην Ολομέλεια σήμερα θα έπρεπε τουλάχιστον να μας απασχολήσει το θέμα. Ο ε, Υπουργός Σαλβίνη ξέρει τις υποχρεώσεις του δυνάμει του διεθνούς δικαίου και Δυστυχώς είδαμε πολλούς μετανάστες οι οποίοι δυστυχώς έχουν παραμείνει χωρίς νερό και τροφή. Είδαμε ε, μία κατάσταση απαράδεκτη. Αυτό δεν είναι θέμα Μάλτας ή Ιταλίας. Μπορούμε να το λύσουμε μόνο με συγκεκριμένη δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς σε αυτή την αίθουσα θα πρέπει να το εξασφαλίσουμε αυτό. Έτσι θα διασφαλίσουμε τις ευρωπαϊκές αξίες. Αποτύχαμε αυτή τη βδομάδα. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε έτσι ώστε να ληφθούν οι δύσκολες αποφάσεις δηλαδή το σύστημα του Δουβλίνου θα πρέπει να αναθεωρηθεί για να υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ όλων των κρατών μελών. Επίσης δεν θα πρέπει να δεχτούμε τη θέση και δράση των διακινητών και θα πρέπει να αντιδράσουμε από πλευράς ε, αντιπροσωπιών όλων των ε, υπηρεσιών μας και γραφείων ανά τον κόσμο. Ε, σήμερα ευτυχώς η Ισπανία ανέλαβε δράση, αλλά αυτό θα ξανασυμβεί και αύριο αν δεν κάνουν κάτι οι πρωθυπουργοί επί του θέματος. Δεν ήθελα να γίνει συζήτηση. Δεν άκουσα αυτά που προείπε η κυρία, αλλά με ενέπνευσαν. Μπορούν να επαναληφθούν. Ηρωνικό σχόλιο. Λοιπόν, τώρα ας ψηφίσουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, λίγη ησυχία. Ήθελε η συνάδελφος να αναφερθεί σε κάτι. Και παρακαλώ δεν θέλω αντιδράσεις ιδιαίτερα από εκείνους που δεν έρχονται στην Επιτροπή Λίμπε συχνά. Η κυρία Μέτσολα έθιξε αυτό το διαδικαστικό γιατί εθίγει στην Ολομέλεια κάτι που δεν προβλεπόταν και θα γίνει μια συζήτηση την Τετάρτη ενώπιον του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις. Υποθέτω ότι πολλά μέλη της Επιτροπής θα συμμετάσχουν στη συζήτηση της Τετάρτης σε σχέση με την κατάσταση στη Μεσόγειο και τις νέες αφήξεις. Σας ευχαριστώ για αυτό το θέμα που θίξατε. Τώρα περνάμε στην ψηφοφορία. Έχουμε δύο ψηφοφορίες. Τώρα, ε, σε σχέση με την προστασία που παρέχεται από την, ε, ως προς την ασπίδα προστασίας η κυρία Μακοβέη. Σήμερα ψηφίζουμε τον κανονισμό της, ε, της του Οργανισμού Ασφάλειας. Αυτό ο οργανισμός θα κάνει τις βάσεις δεδομένων διαλειτουργικές. Δεν ήταν αποτελεσματικό μέχρι στιγμή στη γενοτών, διότι ψάχναμε ε, δεδομένα σε 10 διαφορετικές βάσεις δεδομένων. Ε, είναι πιο εύκολο να τις βρίσκουμε τις ε, πληροφορίες μόνο μιας και να κάνουμε μια σωστή και αποτελεσματική ανάλυση των δεδομένων. Σήμερα μπορούμε να δουλεύουμε συντονισμένα, με ταχύτητα και να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία και την πραγματικότητα Ευχαριστώ τους ε, συναδέλφους με τους οποίους διανύσαμε ένα μεγάλο ταξίδι, αλλά φτάσαμε αισίως στο τέλος αυτού του ταξιδιού. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ λοιπόν να ψηφίσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Has Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 47 υπέρ, 4 κατά και 6 αποχές. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Και τώρα περνάμε στη δεύτερη ε, ψηφοφορία επάρκεια προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΑ. Η κυρία Γκρίσμπεκ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Κλοντ. Για αυτήν την ψηφοφορία οι φιλελεύθεροι θα ήθελαν στην τροπολογία 87 της Σοφή Ίνφελτ να προσθέσουμε κάτι. Στην αρχή δηλαδή της τροπολογίας 87 να προσθεθεί το εξής. Πιστεύω ότι έχετε τη διατύπωση, είναι το 24α στα αγγλικά consider that Δηλαδή ε, η φράση ουσιαστικά αναφέρεται στη συμμόρφωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Σεπτεμβρίου του 2018. Ευχαριστώ πολύ. Πρόκειται για προφορική ε, τροπολογία. Είναι επιπρόσθετη προστίκη μάλλον στην ε, 87 ε, ε, δηλαδή ε, εάν δεν αντιδράσει η ΕΠΑ και δεν δεχτεί αυτές τις προτάσεις μέχρι το Σεπτέμβριο του 18, θα πρέπει να λήξει η ασπίδα προστασίας που παρέχεται έναντι των ΕΠΑ. Έχει κανείς αντίρρηση? Όχι. Ωραία. Θα ψηφίσουμε όταν φτάσουμε σε αυτή την τροπολογία. Ευχαριστούμε Νάταλη. Λοιπόν τώρα αρχίζει η ψηφοφορία η Ρομπέρτα. Λυπάμαι που επανέρχομαι και κατανοώ ότι αυτή η προφορική τροπολογία ήθελε να γεφυρώσει τις διαφορές της πολιτικές ομάδες, όμως για διαδικαστικούς λόγους και για τους λόγους που εξήγησα στο email που σας έστειλα την προηγούμενη εβδομάδα πιστεύουμε ότι υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω διαπραγματεύσεων και θα θέλαμε να δούμε ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα αν μπορέσουμε να ζητήσουμε ε, αναβολή της ψηφοφορίας. Για να διασαφηνίσω το θέμα προς τους συναδέλφους, η κυρία Μετσόλα ε, εκ μέρους του ΕΛΚ στις 9 Ιουνίου ε, ζήτησε να αναβληθεί η ψηφοφορία. Θα πρέπει να ψηφίσουμε δυνάμει του άρθρου 119 του εσωτερικού κανονισμού εδώ, ενώπιον της Επιτροπής. Θα σας διαβάσω λοιπόν, εάν ε, δεν φτάσουμε σε ένα ε, κατόφλι ψήφων για την αναβολή, τότε, ε, θα, τότε θα γίνει η ψηφοφορία για να αποφασίσουμε κατά πόσο μπορεί να γίνει αναβολή με απλή πλειοψηφία. Αν ψηφίσετε ναι, είσαστε υπέρ της αναβολής. Αν ψηφίσετε όχι, σημαίνει ότι δεν γίνεται αναβολή της ψηφοφορίας. Αν ψηφίσετε ναι, ε, πράσινο σημαίνει ότι δέχεστε την αναβολή. Αν ψηφίσετε όχι, κόκκινο σημαίνει ότι δεν αναβάλλεται η ψηφοφορία. Λοιπόν, αν θέλετε να γίνει η ψηφοφορία, κόκκινο. Αν δεν θέλετε και θέλετε να αναβληθεί, πράσινο. Θέλετε να το επαναλάβω για τέταρτη φορά. Εντάξει, ας ψηφίσουμε. Για την ενδεχόμενη αναβολή άρχεται. Πέρας. Άρα γίνεται η ψηφοφορία. Για ευνόητους λόγους το επανέλαβα τέσσερις φορές. Αν κάνατε λάθος, είναι πολύ αργά. Λοιπόν, ας ψηφίσουμε. Αρχίζει ψηφοφορία. Η 20 άρχεται η ψηφοφορία. Okay, colleagues, can we pause for one minute? The SND have one member too many, so one member. Ένας υπεράριθμος από τους σοσιαλιστές. Να αποσυρθεί μια κάρτα παρακαλώ. Uh, no, I have just got confirmation uh, from the secretary that wasn't. Έχω επιβεβαίωση από τη γραμματεία. Ωραία, αποσύρθηκε μία ψήφος. Πέρας και εγκρίνεται. 22. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Παραμένει ανοιχτή. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 28, πρώτο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 30. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 31. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 35. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 36. Πρώτο τμήμα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 38. Πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 40. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 41. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 42 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 46 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 47 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 48 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 52 άρχεται. 52. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 56. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 57. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 58. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 59. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 65. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 66. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 67. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 68. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 69 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 74 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 75. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 76. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 77. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 78. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 80. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 79 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 82 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται συμβαστική 7 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται. Α, τώρα περνάμε στην προφορική 87, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 87. Άρχεται η ψηφοφορία. Μα αυτή δεν ψηφίσαμε τώρα. Ζητώ συγγνώμη, 87, 88 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα πάμε στα έχοντας υπόψη συμβαστική 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 9 στέγοντας υπόψη άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται τροπολογία 6 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται τροπολογία 7 άρχεται η ψηφοφορία πέρας Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται. 11 άρχεται πέρας απορρίπτεται 12 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 13 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 15 ε, η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 16 η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 17 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 18 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται τροπολογία 19 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται και ψηφίζουμε το τελικό κείμενο όπως έχει διαμορφωθεί με ονομαστική ψηφοφορία η οποία και αρχίζει Πέρας. 29 ε, υπέρ 25 κατά, τρεις αποχές, άρα εγκρίνεται. Και τελειώσαμε με την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ πολύ. Um, Συνάδελφοι, εάν θέλετε να παραμείνετε στη συνεδρίαση, παρακαλώ λίγη τάξη. Ο Επίτροπος Κίνγκ είναι μαζί μας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με τα υπόλοιπα θέματα στη μερίσια διάταξη. Αν θέλετε να αποχωρήσετε, αποχωρήστε με ησυχία. Σας ευχαριστώ. So, um, Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συναδέλφους που είναι μαζί μας για αυτό το θέμα της μερίσιας διάταξης. Ξέρω ότι μερικοί δυσκολευτήκατε πάρα πολύ, είχατε φρικτό ταξίδι μέχρι να φτάσετε εδώ, ε, πολλές ώρες στα τρένα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ, δεν είναι εύκολο, Δευτέρα βράδυ και ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Επίτροπο Κίνγκ που είναι εδώ. Ξέρω ότι η Δευτέρα στα Στρασβούργο ε, δεν είναι και καλύτερη ημέρα, αλλά έχουμε αυτή τη συζήτηση που διευθετήθηκε για σήμερα, όπως γνωρίζετε. Είναι η, η έκθεση προόδου της Ένωσης Ασφάλειας θα ήθελα να πω ότι στις 17 Απριλίου εισαγωγικά θα έλεγα η Επιτροπή ε, ξέδωσε την 14η έκθεση προόδου ε, μαζί με νομοθετικές ε, προτάσεις για τη διευκάλυση της διασυνοριακής πρόσβασης σε πληροφορίες στις ε, αρχές επιβολής του νόμου ε, διάφορα έγγραφα που μπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση των κανόνων για τις πρόδρομες ουσίες συγκρατικών και τις αγωγές των πυρομαχικών όπλων και είμαστε με τον Επίτροπο εδώ, ο θα μας αναλύσει αυτό το πακέτο και η Νάταλη που είναι επικεφαλής της, επικεφαλής της Επίτροπης ΤΕΡ που βρίσκεται σήμερα εδώ επίσης. Ο Επίτροπος King ε, Θα πρέπει να μιλήσω για το νομοθετικό πακέτο. Είχα και μερικά άλλα πράγματα. Νομίζω είναι καλύτερα όμως να δώσουμε το λόγο στον Επίτροπο, ε, γιατί τώρα έχετε την ε, πλήρη προσοχή των συναδέλφων. Ξέρω ότι είναι δύσκολη ώρα, είναι κουρασμένοι οι συνάδελφοι, είχαν φρικατό ταξίδι μέχρι να φτάσουν εδώ. Κάποια από τα μέλη του προσωπικού μου ακόμη είναι στο τρένο και αντιλαμβάνουμε πόσο δύσκολο είναι για σας. Επίτροπε, ε, σας καλωσορίζουμε. Ας ακούσουμε την σύνοψή σας και μετά μπορούμε να κάνουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ και πάλι που βρίσκεστε εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αξιότιμα μέλη, συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ που ε, ε, έχετε ξεκινήσει ένα διάλογο σε αυτά τα θέματα. Πριν από μερικέ εβδομάδε είχαμε προτείνει την τελευταία έκθεση πρόοδου με το πακέτο μέτρων που θα συζητήσουμε τώρα. Ενδεχομένω με αυτή την ευκαιρία να πω και μερικά λόγια σχετικά με την επόμενη έκθεση της ε, Ένωσης Ασφάλειας που θα εκδοθεί αυτή τη βδομάδα και που σημειώνει πρόοδο σε κάποιους τομείς. Το πακέτο Απριλίου, το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα, ε, μπαίνει στη καρδιά της δουλειάς μας ε, στην Ένωση Ασφάλειας ε, για να κλείσουμε το χώρο στον οποίο λειτουργούν οι εγκληματίες και οι τρομοκράτες για να δυσχεραίνουμε το έργο τους στο προγραμματισμό επιθέσεων. Το πακέτο των προτάσεων που συζητάμε εδώ είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να δυσκολεύει ε, την διακίνηση των τρομοκρατών, το, τη χρηματοδότησή τους, ε, το να βρουν εκρηκτικά και αντιμετωπίσουν ε, εμπόδια στο, στο έργο που, που κάνουν. Με τις εκλογές που επικίνδυνται του χρόνου, ελπίζουμε να συνεργαστούμε αποτελεσματικά έτσι ώστε να έχουμε αποτελέσματα στις πλήστες από αυτές τις προτάσεις στον χρόνο που μας απομένει. Εάν θέλετε μπορώ να μιλήσω για κάποιες πρωτοβουλίες. Πρώτα απ' όλα και με καμιά σειρά προτεραιότητα ένα θέμα σημαντικό είναι προτάσει για την βελτίωση της προσβασής στην ηλεκτρονική, ε, στα ηλεκτρονικά στοιχεία. Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο, χρονοβόρο. Μερικές φορές ε, είναι πολύ αργή αυτή η διαδικασία, ιδιαίτερα όταν ε, τα στοιχεία βρίσκονται σε διαφορετικές δικαιοδοσίες. Για να μειώσουμε λοιπόν τις καθυστερήσεις στην εξασφάλιση αποδεικτικών ψυχίων συνοριακά, έχουμε δύο νομοθετικές πρότασεις, έναν κανονισμό και μια οδηγία που θα παρέχουν στις αρχές επιβολής του νόμου κάποια νέα εργαλεία για να εξασφαλίζουν αποδεικτικά στοιχεία email, κείμενα, whatsapp, ε, ε, μηνύματα, messenger για τη διερεύνηση και την δίωξη εγκλημάτων συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας και του εγκλήματος των κυβερνοχώρων. Ε, τα μέτρα περιλαμβάνουν τη δυνατότητα των δικαστικών αρχών, όχι της αστυνομίας, των δικαστικών αρχών να ζητάνε κατευθείαν από τους παρόχους ε, υπηρεσιών από μια άλλη δικαιοδοσία να παρέχουν ε, τα αποδεικτικά στοιχεία. Οποιοςδήποτε πάροχος που παρέχει υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει την υποχρέωση να απαντάει σε αυτό το αίτημα και υπάρχουν χρονοδιαγράμματα που καθορίζονται και ο στόχος είναι να υπάρχει ανταπόκριση εντός 10 ημερών κατά όρο και με ταχύτητα σε εντός ορισμένων ορών σε κάποιες επίγουσες περιπτώσεις. Οι πάροχοι ε, πρέπει να διατηρούν ορισμένα στοιχεία με την χρήση της εντολής διατήρησης. Αυτές ε, οι εντολές χρησιμοποιούνται μόνο στη διαδικασία δικαστικών διαδικασιών και ε, εφαρμόζονται όλες οι εγγύησεις. Ε, δεδομένης της φύσης αυτών των εντολών, των διαταγών, έχουμε τις ε, εγγύσεις που εφαρμόζονται στους παρόχους υπηρεσιών. Έχουμε και κάποια πρακτικά μέτρα για να απλωσεύσουμε τις ε, διαδικασίες ανάμεσα στις δικαστικές αρχές και τις αρχές επιβολής του νόμου και τους παρόχους υπηρεσιών γύρω από τα υφιστάμενα εργαλεία. Σε αυτή τη διαδικασία γνωρίζουμε ότι δεν ε, αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα σε κενό. Υπάρχουν εξελίξεις σε άλλα μέρη του κόσμου που η έγκριση του Cloud Act στην Αμερική, του νόμου Cloud. Πιστεύουμε ότι οι προτάσει μας αποτελούν μια βάση για μια συνεκτική προσέγγιση τόσο εντό τη ευρωπαϊκή Ένωσης όσο και από την Ευρωπαϊκή ε, ε, Ένωση σε διεθνέ επίπεδο λαμβανομένων υπόψη των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωση και των ε, εγγυήσεων όπως ε, του δικαιώματος ε, ενδίκων μέσων. Ένα δεύτερο θέμα το οποίο εξετάσαμε ήταν η, η πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές πληροφορίες σε εξέλιξη είναι αυτό το θέμα. Είναι εύκολο για τους εγκληματίες και τους τρομοκράτες να δρουν σε διάφορα κράτη-μέλη και να ε, μεταφέρουν χρηματικά ποσά. Ε, οι αρχές επιβολής του νόμου πρέπει να έχουν ρυθισμένη πρόσβαση σε χρηματοοικονομικά στοιχεία για να κατοπελμούν το σοβαρό έγκλημα. Η δεύτερη πρόταση λοιπόν στοχεύει στη διευκόλυση αυτή τη πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία και η προτενόμενη οδηγία θα δώσει στι αρχέ επιβολή του νόμου ε, την πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία που χρειάζονται για τη διαρρεύνησή του, χωρί να ζητάνε γενικές, γενικά αιτήματα σε όλου του χρηματοπιστωτικού οργανισμού, γιατί αυτό είναι χρονοβόρο, μη αποτελεσματικό και βέβαια ε, ενέχει κινδύνους διότι απευθύνεται σε περισσότερα άτομα από ό,τι θα έπρεπε. Ε, θα παρέχει στις ε, αρχές, στις αρχές άμεση πρόσβαση στα στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται στα Εθνικά Κεντρικά Μητρώα των Τραπεζικών Λογαριασμών. Αυτή η οδηγία θα ενισχύει τη συνεργασία ανάμεσα στα, στις αρχές πληροφοριών και τις αρχές επιβολής του νόμου των κατών μελών, καθώς και με την Ευρωπόλ. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε αυτές τις αρχές να ετούνται ε, αυτών των πληροφοριών. Ε, η πρόταση επίσης προβλέπει ε, εγγύησεις και διασφαλίσεις ό,τι αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ένα άλλο τομέα που εξετάσαμε ήταν η βελτίωση των ε, στοιχείων ασφάλειας σε θέματα δελτίων ταυτότητας. Ε, τα στοιχεία ταυτότητας και η παραποίηση είναι θέμα ανησυχίας, διότι επιτρέπει στους εγκληματίες και τους τρομοκράτες να ε, εισέλθουν στην Ένωση και να διακινηθούν χρησιμοποιώντας παραποιημένα στοιχεία. Κάπου 18 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή έχουν ε, δελτία ταυτότητας που δεν ε, διαβάζονται, που δεν έχουν βιομετρικά στοιχεία. Και αυτό ε, δημιουργεί πρόβλημα. Για να το αντιμετωπίσουμε αυτό, η Επιτροπή πρότεινε βελτιώσεις στη, στην χρήση των δελτιών ταυτότητας και σε, στα έγγραφα διαμονής. Δεν προτείνουμε ε, μια ευρωπαϊκή, ένα ευρωπαϊκό δελτίο ταυτότητας. Ο στόχος ε, θα είναι να δημιουργήσουμε κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χρησιμοποιώντα τα βιομετρικά στοιχεία, ε, δαχτυλικά αποτυπώματα, να είναι υποχρεωτικά στις χώρες που ήδη εκδίδουν εθνικά δελτία ταυτότητας. θα υπάρχουν βέβαια ισχυρέ εγγύσει και δικλείδες ασφαλείας. Θα ήθελα να τονίσω ότι δεν γίνεται υποχρεωτική εισαγωγή των δελτίων ταυτότητας σε χώρες που δεν τα τα έχουν, αλλά ενισχύει και αναβαθμίζει τα συστήματα σε χώρες που υπάρχουν τα δελτία ταυτότητας και δίνεται χρόνο στις χώρες για να εκδοθούν νέες ε, ταυτότητες. Ένας άλλος τομέας ήταν οι πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών, ένα κοινό θέμα. Ε, που γνωρίζουμε ε, ε, είναι η χρήση των αυτοσχέδιων εκρηκτικών. Χρησιμοποιούνται με πρόδρομες ουσίες που είναι εμπορικώς διαθέσιμες. Αυτή τη στιγμή κράτη-μέλη έχουν διαφορετικά καθεστώτα σχετικά με αυτά στις πρόδρομες ουσίες που δεν είναι ιδανικά. Πρέπει να κλείσουμε αυτό το θέμα. Ήταν θέμα που η Επιτροπή προτείνει την αναθεώρηση του εφαστάμενου κανονισμού για τις πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών, ενισχύοντας και ε, ε, τους κανόνες για να κλείσουμε κάποια κενά και για να σταματήσει η κατάχρηση ε, των πρόδρομων ουσιών. Ο Στόχος είναι η απαγόρευση κάποιων εκρηκτικών και πρόδρομων ουσιών που χρησιμοποιούνται για την ε, παρασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών. Οι κράτη-μέλη θα πρέπει να ε, ε, κατέχουν άδειε για την κατοχή αυτών των πρόδρομων ουσιών και ε, θα πρέπει να λαμβάνονται αρκετά στοιχεία υπόψη κατά την χορήγηση αυτών των αδειών. Κάτι άλλο ήταν η ενίσχυση των ελέγχων ε, για την εισαγωγή και την εξαγωγή όπλων. Έχουμε λάβει ορισμένα μέτρα, αρκετά μέτρα όπως έχουμε συζητήσει, για τον περιορισμό της προμήθειας πυροβολών όπλων ενισχύοντας διάφορα μέτρα. Αυτή η πρόταση τώρα ενισχύει ε, τους κανόνες για την εισαγωγή και εξαγωγή των πυροβολών όπλων. Έχουμε εκδώσει μια σύσταση που βελτιώνει τις διαδικασίες ελέγχου και απαιτεί από τα κράτη-μέλη να έχουν ε, συστηματικούς ελέγχους στοιχείων όλων των ατόμων που αιτούνται, ε, αδειών εξαγωγής. Αυτές είναι σημαντικές προτάσεις. Όπως είπα και εξ αρχής, ε, προσβλέπουμε την άνοιξη του διαλόγου μαζί σας ε, άμεσα στα θέματα που θέλουμε να προχωρήσουμε, έτσι ώστε να πετύχουμε αποτελέσματα το συντομότερο δυνατόν πριν από το πέρας αυτής της θητείας. Με στη διάθεση των εισηγητών, της κυρία Σίπελ, του κύριου Μεμακίνς, του κύριου Ντιπρέ και του κύριου Ραντεύ και προσβλέπω στη συνεργασία μας για να ε, εξετάσουμε αυτά τα θέματα. Και τέλος, αφού έχω το λόγο, αν μου επιτρέπετε, αν θα μπορούσα να ε, δούμε ε, την, την 15η έκθεση πρόοδου της Ένωσης Ασφάλειας που εκδίδεται αυτή τη βδομάδα. Αυτή η έκθεση θα εξετάσει την πρόοδο που έχει επιτελεστεί στην υλοποίηση του σχεδίου δράσης σε για τα χημικά, βιολογικά, ραδιολογικά και πυρηνικά ε, της πυρηνικές απειλές. Δυστυχώς ε, η πρόσφατη επίθεση στο Σάλσμπουρι ε, υπογράμμισε ότι η ετοιμότητα να αντιμετωπίσουμε αυτές τις απειλές δεν είναι πια θεωρητική, είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Προσπαθούμε να μειώσουμε την προσβασιμότητα σε αυτά τα υλικά, να βελτιώσουμε την ετοιμότητά μας, την ανθεκτικότητά μας και να βελτιώσουμε την διεθνή συνεργασία κατά αυτής της απειλής. Επίσης, ε, προτείνουμε να λάβουμε συγκεκριμένα μέτρα κατά του χημικού κινδύνου. Η έκθεση εξετάζει την πρόοδο στην αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου ε, διαδικτυακά από την σύσταση που είχαμε εκδώσει την 1η Μαρτίου και αυτό ε, ακολουθεί την τελική έκθεση της ε, ομάδας εμπειρογνωμόνων για τη ριζοσπαστικοποίηση. Ταυτόχρονα έχουμε κάποιες βραχυπρόθεσμες δράσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των επιβατών σιδηροδρόμων και επίσης ε, για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών. Επίσης άλλα θέματα περιλαμβάνουν την διαλειτουργικότητα που θα την εξετάσουμε αργότερα, την υλοποίηση ε, της οδηγίας για τα στοιχεία των επιβατών και για ε, το, το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και τον, τους κανόνες για την εισαγωγή, εξαγωγή όπλων και είμαι στη διάθεσή σας να συζητήσουμε και για αυτές τις προτάσεις ε, λεπτομερέστερα όταν εκδοθεί η έκθεση ε, και σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε στα θέματα που έχω αναφέρει. Ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε. Έχουμε ένα κατάλογο ομιλητών. Η Ρομπέρτα όλα εκ μέρους του ΕΛΚ. Εγώ ουσιαστικά εκπροσωπώ τον κύριο Ράντερ Μπορώ να δέσω λοιπόν εκ μέρους του όσον αφορά τη θέση, τελική θέση του ΕΛΚ, όσον αφορά τη χρηματοδότηση το, της τρομοκρατίας, βεβαίως και πρόκειται για μία από τις προτεραιότητες του 2015 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό φαίνεται από διάφορα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχει σαφώς ε, εντοπιστεί το θέμα της βελτίωσης στον τομέα της ανταλλαγής πληροφοριών, καλύτερης συνεργασίας ε, σε θέση με τη χρήση όπλων και εγκρικτικών. Η πρόταση που συζητούμε σήμερα, που αφορά ουσιαστικά την χρήση οικονομικών πληροφοριών για την καλύτερη πρόληψη, διερεύνηση και δίωξη τέτοιων ε, πράξεων, Σαφώς χρειάζεται πιο ταχεία συνεργασία, βελτιωμένη συνεργασία. Πρέπει να καλύψουμε τα κενά που υπάρχουν σήμερα στην υπάρχουσα νομοθεσία, καθώς και τις διατάξεις οι οποίες ισχύουν για να γίνει πιο ισχυρό το οικοδόμημα αντιμετώπιση αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα που έχει θίξει πάρα πολλές φορές η Eurocall, που είναι η νομοποίηση παρανομών κονδυλίων. Το θέμα της ε, διαφάνειας για τους καταπολέμησης διαφοράς είναι κάτι που σαφώς θα πρέπει να ενισχυθεί επίσης. Είναι κάτι που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και θα πρέπει να τηρηθεί η αρχή της αναλογικότητας. Χρειάζονται επικοδομητικές συζητήσεις με τους κοιόδης και βεβαίως ελπίζουμε να ολοκληρωθεί η συζήτηση και η διαδικασία με την Επιτροπή πριν το τέλος ε, του επόμενου χρόνου. Ευχαριστώ πολύ. Καλύψατε και το κύριο Ράντεφ, η Μπίργκιτ Σίβολ. Είναι συντονίστρια για την ομάδα των σοσιαλιστών. Ευχαριστώ πολύ, Κλοντ. Με μεγάλη χαρά έχουμε ανταλλαγή απόψη για θέματα ασφάλειας με τον Επίτροπο Κίνγκ. Πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της ασφάλειας για τους πολίτες. Εκπλήσωμε, διότι συνήθως τα θέματα της ασφάλειας συζητώνται σε πολύ περιορισμένο πλαίσιο. Μιλάμε για την προστασία των πολιτών κατά των εγκληματιών, αλλά και θα πρέπει να προστατεύσουμε και την ελευθερία έκφρασης. Κύριε Κίνγκ, ζητώ συγγνώμη, αλλά θα ήθελα να το αναφέρω αυτό. Λυπούμε διότι δεν υπάρχει καμία πρόοδο σε θέματα όπως προστασία των προσωπικών δεδομένων, το λεγόμενο e-privacy. Ακούσαμε την δέσμευση, προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των επικοινωνιών των πολιτών μας. Θα πρέπει να νιώθουν ασφαλείς, όπως ακριβώς προστατεύουμε δηλαδή την εγκληματικότητα. Διάβασα προσεκτικά τις προτάσεις σας, τα θέματα που επεξεργάζεστε, το θέμα των ηλεκτρονικών στοιχείων και βεβαίως υπάρχουν πάντα πολύ σοβαρά ερωτήματα για τόσο σοβαρά θέματα. Έχω λοιπόν ε, ερωτήσεις. Δεν θέλω να μπω στην ουσία. Η ερώτησή μου είναι αν για όλες τις πολιτικές ομάδες το θέμα αυτό είναι τόσο σημαντικό. Την προηγούμενη εβδομάδα άκουσα ότι δεν υπάρχουν σκιώδεις για όλες τις πολιτικές ομάδες. Δεν έχουν διοριστεί ακόμα. Με ενδιαφέρει να δω πώς θα εξελιχθεί αυτό το θέμα. Μιλήσατε για το Κλάντεκ και εδώ έχουμε ερωτήσεις, αναπάντητες. Μιλήσατε και για τις ασφαλιστικές δικλίδες τις εγγύησει, τι ακριβώς είναι αυτές και τι προτείνεται έτσι ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν αυτές τις εγγύησεις και τις ασφαλιστικές δικλείδες άμεσα, όχι στην τελευταία φάση της διαδικασίας. Ανησυχούμε λοιπόν ε, όσον αφορά τη λειτουργία αυτών και χρειάζεται συνεργασία με νομικούς, με φορείς παραχής υπηρεσιών και αυτό που κυρίως πρέπει να διασφαλίσουμε είναι την ελευθερία και την προστασία, την ασφάλεια των πολιτών μας. Το θέμα των ε, ταυτοτήτων, το θέμα των ε, αδειών παραμονής, Ξέρετε, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, άκουσα προσεκτικά αυτά που είπατε. Θα περιοριστώ στην έκθεση, η οποία αφορά τα δικά μου θέματα, δηλαδή στοιχεία ασφάλειας στα δελτία ταυτότητας. Χαιρετίζω αυτή την πρωτοβουλία για δύο διαφορετικούς μεταξύ τους λόγους. Πρώτον, το θέμα της ασφάλειας. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι πιστεύω ότι πρέπει να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία όλων και η δουλειά όλων. Η μελέτη αντικτύπου, η οποία έγινε πριν υποβληθεί αυτή η πρόταση, αναφέρει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν 250 διαφορετικά έντυπα που αφορούν τα δελτία ταυτότητας και τις άδειε παραμονής. Μα πώς είναι δυνατό να το συνεχίζουμε αυτό και να το δεχόμαστε. Η απλοποίηση για όλους τους πολίτες είναι απαραίτητη. Ακόμα και για αυτούς που πρέπει να διαβάσουν, να κατανοήσουν και να ελέγξουν αυτά τα έγγραφα ταυτότητας. Για τη διευκόλυνση λοιπόν και της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών αλλά και του ελέγχου των εγγράφων αυτών είναι απαραίτητη η απλοποίηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θα ήθελα επίσης να πω ότι έξυπνα η Επιτροπή πρότεινε πρώτον μία μη υπερβολική πρόταση, δηλαδή δεν επιβάλλει στα κράτη-μέλη που δεν έχουν ε, ταυτότητα να δημιουργήσουν. Μόνο αυτοί που έχουν δελτία ταυτότητες θα πρέπει να υιοθετήσουν τον, τη νέα μορφή της με, τις, με τα νέα στοιχεία ασφάλειας. Δεύτερο, και αυτό πρέπει να διευκρινιστεί, δεν θα δημιουργήσουμε έναν ε, Big Brother με όλα αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή, δεν θα υποχρεώσουμε τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν μια κεντρική βάση δεδομένων με όλα αυτά τα στοιχεία. Δεν θα ενσωματωθούν δηλαδή τα στοιχεία ταυτότητας όλων των Ευρωπαίων πολιτών σε ένα κεντρικό σύστημα τύπου Big Brother. Αυτό είναι πάρα πολύ ουσιαστικό και πρέπει να το επαναλάβουμε. Η πρόταση της Επιτροπής, ναι βλέπω ότι ο χρόνος τρέχει. Πρόκειται για στοιχεία που αφορούν τα δακτυλικά αποτυπώματα και άλλα βιολογικά στοιχεία. η ανήλικοι. Πρέπει να προστατεύσουμε τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό που προστατεύουμε τους μετανάστες. Δεύτερον, η διάρκεια των νέων αυτών εγγράφων. Το κόστος είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να αξιολογηθεί για τη δημιουργία αυτών των νέων δελτίων ταυτότητας. Πιστεύω ότι οι δύο προτάσεις της Επιτροπής πρέπει να υποστηριχθούν από την Επιτροπή μας και από το Κοινοβούλιο γενικότερα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος να σας υπενθυμίσω ότι οι διερμηνείς σήμερα δεν θα υπερβούν τον χρόνο εργασίας τους. Σας παρακαλώ πολύ λοιπόν τηρείτε το χρόνο μιλία σας, εάν μπορείτε. Επανέρχομαι στον κατάλογο μιλητών η Ναταλή Γκρίσπεκ, η οποία είναι επικεφαλής Αρμόδης επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Επίτροπο Julian King που είναι εδώ για να συζητήσουμε θέματα προστασίας και θέματα ισορροπημένης προσέγγισης για τους Ευρωπαίους πολίτες. Υπάρχουν πολλές και ενδιαφέρουσες προτάσεις που αφορούν τους στόχους συνεργασίας, ανταλλαγή πληροφοριών, καταπολέμηση της ε, τρομοκρατίας, αντιμετώπιση των τρομοκρατών, παρακολούθηση των τρομοκρατών, της χρηματοδότησης επίσης της τρομοκρατίας. Πολύ σύντομα λοιπόν θέλω να μιλήσω για τις πρόδρομες ουσίες για τη δημιουργία εκρηκτικών. Η πρόταση για το θέμα αυτό μου φαίνεται ότι θα μας επιτρέψει να δημιουργήσουμε ένα πιο αποτελεσματικό εργαλείο και ότι πραγματικά λαμβάνει υπόψη τας όλα τα νέα δεδομένα για τη δημιουργία αυτών των εκρητικών ε, υλών με τρόπο που θα μπορούσε να βοηθήσει πρόχειρες ε, τρομοκρατικές επιθέσεις, τρομοκρατικές επιθέσεις χαμηλού κόστους να πολλαπλασιαστούν. Χρειάζονται λοιπόν εδώ σίγουρα καλύτεροι ορισμοί των ενιών. Πρέπει να βασιστούμε σε πιο σαφείς ορισμούς των χρηστών και όπως ξέρετε οι αλυσίδες για τη δημιουργία αυτών των προϊόντων και υλικών μπορεί να είναι πολύ σύντομες ή πάρα πολύ μεγάλες και θα πρέπει να καλύψουμε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Οι ορισμοί λοιπόν, έτσι ώστε τα άτομα, οι μικρομεσές επιχειρήσεις, οι μεγάλες επιχειρήσεις, η δημόσια διοίκηση, θα πρέπει να μπορούν να εντοπίσουν, να γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται. Δεύτερο, χρειάζεται εναρμόνιση. Τα κράτη-μέλη δεν χρησιμοποιούν τον ίδιο τρόπο αδειοδότησης και αυτό σίγουρα μπορεί να έχει επιπτώσεις όσον αφορά την υλοποίηση και την αποτελεσματικότητα αυτού του κανονισμού. Ευχαριστώ. Κύριος Μάνκινς, θέλετε να πάρετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω λετονικά, αν μπορώ. Σε σχέση με τις ε, πρόδρομες εκρηκτικές ουσίες, είναι πολύ καλό για το ότι η Επιτροπή θα αλλάξει τον κανονισμό 98 κάθετος 2013 και ιδιαίτερα σε σχέση με την αδειοδότηση και καταγραφή. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα μητρώων όπως τη... Γαλλία. Στη χώρα μου και στην Εστονία υπάρχει απαγόρευση. Θυμάμαι ότι στα παιδικά μου χρόνια μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε ε, διάφορες ουσίες για να κάνουμε ε, μικροβομβίδια. Ε, Ένα συμμαθητής μου έχασε το δάχτυλό του και μπορεί κανείς να κάνει μία πρόσμιξη και είναι έτοιμη μία εκρηκτική ουσία. Και κάτι άλλο. Αφορά την χρήση χόρτου στην Ολλανδία. Μπορεί κανείς να αγοράσει χόρτο, μαριχουάνα δηλαδή, στην Ολλανδία και να την καπνίσει στην Εστονία ή στη Λετωνία. Γι' αυτό θα πρέπει να το δούμε συνολικά το όλο ζήτημα. Πώς το βλέπετε. Δεν θα ήθελα να σας πω ότι γίνεται στη Γλασκόβη, ας το αφήσουμε αυτό το θέμα. Χαίρομαι που ήσασταν σαφείς. Coordinators, Cornelia Ernst, please, Cornelia. Ja. <laughs> Also, ja, Aussprache über das Sicherheitssystem. Κοιτάξτε, εδώ αναφερόμαστε στο πακέτο που αφορά την ασφάλεια. Και πολύ ήρεμα μπορώ να σας πω ότι δύσκολα μπορώ να τα συμπεριλάβω όλα αυτά σε ένα κείμενο. Τώρα μιλάμε για τις εκρηκτικές ύλε. Κοιτάξτε, ουσιαστικά η εσωτερική λογική η οποία πρέπει να διατηρηθεί για έναν απλό άνθρωπο δεν είναι εύκολο διαβάζοντας τις προτάσεις αυτές. Το λέω με κάθε, αν θέλετε, βίκια. Για το πρώτο λοιπόν σημείο, όταν μιλάμε για αποδεικτικά στοιχεία, θα νομίζω θα πρέπει να ξαναδούμε τη διατύπωση. Βασικά, ναι, θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε λίγο τις προτάσεις αυτές, να τις συμπληρώσουμε και να επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Συμφωνούμε με αυτό. Απλοποίηση και επιτάχυνση. Υπάρχουν παρόλα αυτά κίνδυνοι και γι' αυτό και θα ήθελα να πω στον Επίτροπο Κίνγκ τα εξής. Πώς μπορούμε να, όταν πρόκειται για προστασία δεδομένων, αν θέλετε, να κάνουμε διάκριση μεταξύ μεταδεδομένων και δεδομένων. Εδώ και οι εισαγγελίε θα πρέπει να έχουν μια πολύ σαφή ε, εικόνα. Δεύτερον, οι ποινές, η διάρκεια των ποινών, το ύψος των ποινών. Ούτε εδώ είναι σαφές αν τηρείται η αναλογικότητα. Και η ερώτηση την οποία την ξέρετε γιατί την έχετε ξανακούσει. Τι εγγύησεις υπάρχουν για τα ενδιαφερόμενα άτομα. Προστασία των δεδομένων, ναι. Προστασία της ιδιωτικής ζωής, ναι. Το θέμα όμως είναι να υπάρχουν εγγύησεις και όσον αφορά τη διαδικασία. Αυτό, αν θέλετε, θα πρέπει να μας το εγγυηθείτε. Ναι, επιταχύνουμε τις διαδικασίες, σωστό, αλλά χρειάζονται κάποιες εγγυήσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Τόμας Τσιντόφσκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε, και για την παρουσία σας. Δεν θα μιλήσω τυπικά και δεν θα σας ευχαριστήσω για όλα όσα έχετε κάνει. Θα μιλήσω επί της ουσίας. Νομίζω ότι η πρότασή σας είναι πολύ σημαντική για την καταπολέμηση της ε, τρομοκρατίας. Το πακέτο είναι πολύ σχηδές και πολύ καλά προετοιμασμένο και νομίζω ότι είναι απόλυτα λογικό. Σε σχέση με τις πρόδρομες εκρηκτικές ε, ύλες, νομίζω ότι όλα αυτά συσχετίζονται με τις ε, επιθέσεις στο Βέλγιο και τη Γαλλία. Ήταν αυτοσχέδιοι οι μηχανισμοί και στις δύο περιπτώσεις, άρα η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν μπορεί να αποτρέψει τις αυτοσχέδιες αυτές βόμβες. Θα πρέπει να δούμε και την ε, πρόσβαση στις πρόδρομες ουσίες, Χτες ε, έλεγξα κατά πόσο εγώ θα μπορούσα να ε, φτιάξω μία αυτοσχέδια βόμβα. Θα μπορούσα να βρω όλα τα υλικά στο ίντερνετ. Ναι, μου χρειάστηκαν τρία λεπτά μόνο για να εντοπίσω τις ε, πρόδρομες ουσίες. Θα πρέπει να ταυτοποιήσουμε αυτούς που τις αγοράζουν όμως. Δηλαδή να ελέγξουμε τις επιγραμμικές πωλήσει και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει και έλεγχος συμμόρφωσης ως προς αυτές τις διατάξεις. Επίσης δεν υπάρχει ε, σωστή, δεν υπάρχει ενσυνειδητότητα. Θα πρέπει να βελτιωθεί η πρόταση και να υπάρχει αυτόματη γνωστοποίηση ενδυνάμει δράσεων και ανταλλαγή δεδομένων μέσα από την εφοδιαστική αλυσίδα, γιατί οι ουσίες είναι ξεχωριστές και μόνο όταν ε, αποτελέσουν, γίνουν μία πρόσμιξη, οδηγούν σε εκρηκτική ύλη. Κύριε Επίτροπε, σε πολλές χώρες οι ανταλλαγές ε, χρηματοπιστωτικών ε, συναλλαγών αποτελούν αντικείμενο μυστικών υπηρεσιών. Πώς μπορεί να υπάρχει συνεργασία μέσω της Europol. Και ως προς την αποδόμηση των ε, όπλων, αυτό είναι θέμα που δεν απολά τη συζήτηση. Ευχαριστώ, Κλόντα. Εγώ θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις στον ε, Επίτροπο αφορά την ασφάλεια των δελτίων ταυτότητας και άλλων τέτοιων εγγράφων. Βεβαίως και κάτι πρέπει να αλλάξει εδώ, βεβαίως χρειάζεται μία εναρμόνιση. Απ' την άλλη υπάρχουν τελείως διαφορετική μορφή εγγράφων αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και αυτό που με ενδιαφέρει είναι αν η άποψη της Επιτροπής είναι να κάνει έναν απολογισμό, αν ξέρει σήμερα ποια είναι τα πλαστά, σε ποσοστό, σε απόλυτους αριθμούς, για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε και να ξέρουμε το κόστος αυτής της αλλαγής, αν θα αξίζει τον κόπο. Δεύτερο, δεύτερη ερώτηση που θέλω να κάνω. Αυτός ο κανονισμός θα αρχίσει να ισχύει και 16 αν θέλετε κράτη-μέλη και οι πολίτες τους θα περάσουν σε μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Εκατομμύρια άνθρωποι θα πρέπει να δώσουν τα δακτυλικά τους αποτυπώματα για να ενσωματωθούν αυτά στα δελτία ταυτότητας. 570 εκατομμύρια πολίτες της Ευρώπης. Αναρωτιέμαι λοιπόν από άποψη προστασίας προσωπικών δεδομένων και οι νομικές, ε, αν θέλετε, συμβουλές που σας έχουν δοθεί για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των προσωπικών δεδομένων καλύπτεται από αυτές τις προτάσεις. Κύριε Επιτρόπη, μπορείτε να μου απαντήσετε σε αυτά τα δύο πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα που σας έκανα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Βίκστρομ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Κλόντ και ευχαριστώ κύριε ε, ε, Επίτροπε που βρίσκεστε εδώ αργά το βράδυ της Δευτέρας στο Στρασβούργο για να συζητήσετε το πακέτο ασφαλείας που είναι ύψη της σημασίας για εμάς και νομίζω ότι θα πρέπει να φτάσουμε σε μια συμφωνία ως προς την διαλειτουργικότητα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ανταλλαγής Πληροφοριών. Η καλύτερη πληροφόρηση είναι καλύτερη και θα πρέπει να δούμε τις τεχνικές και πολιτικές προκλήσεις. Τα περισσότερα συστήματα που θα ενταχθούν στη διαλειτουργικότητα βρίσκονται υπό αναθεώρηση και αυτό δημιουργεί σειρά προβλημάτων και οι προτάσεις προσθέτουν ένα στρώμα πολυπλοκότητα σε σχέση με τα προϋπάρχοντα συστήματα. Όπως είδαμε πρόσφατα, η παραβίαση δεδομένων μπορεί να βλάψει ένα πολύ μεγάλο αριθμό πολιτών. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχουν οι σωστές ε, δικλείδες ασφαλείας και αναφερθήκατε σε αυτές ώστε να μην ε, γίνονται αυτές η, να μην υπάρχει αυτή η ρήξη στα συστήματα πληροφόρησης. Πολλές φορές δεν λαμβάνουμε υπόψη τι κάνει η ΦΡΑ, η Επιτροπή Θέμελιδων Δικαιωμάτων και νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τι έχουν εκφράσει. Ε, πρόκειται για τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ευρώπης. Και με βάση αυτά που προελέχθησαν σε σχέση με τον έλεγχο του χώρου Σέγγεν υπήρξαν πολύ μεγάλες ελλείψεις σε σχέση με το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών Σέγγεν. Τώρα, μέσα στα πλαίσια αυτής της διαλειτουργικότητας ε, θα μπορούσαν να υπάρχουν σοβαρές συνέπειες όχι μόνο για τους Ευρωπαίους πολίτες αλλά και για τους πολίτες τρίτων χωρών. Γι' αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω τι προτίθεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε έμπρακτα να υπάρχουν αυτές οι δικλίδες ασφαλείας. Τι σημαίνουν και πώς θα πρέπει να τις ακολουθήσει κάθε κράτος μέλος και να συμμορφώνεται. Γιατί ξέρουμε ότι αυτό είναι το αδύναμο σημείο. Η εφαρμογή και η δέσμευση των κρατών μελών. Σας ευχαριστώ πολύ για την εξαιρετική αυτή συνεργασία, η οποία ελπίζω ότι θα ε, συνεχιστεί. Η κυρία Μποτίλ Βαλέρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα χρειαστεί να βάλετε τα ακουστικά σας αυτή τη φορά. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα πολύ χρήσιμα εισαγωγικά σχόλια. Θα ήθελα να ακούσω πολλά περισσότερα, αλλά νομίζω ότι στο μέλλον θα έχουμε τη δυνατότητα για περαιτέρω πληροφόρηση. Αναφερθήκατε στα μικρά και ελαφρά όπλα. Ε, είμαι σκιώδης, όχι σε όλα αυτά τα θέματα, αλλά ε, είμαι σκιώδης ως προς τις ε, πρόδρομες ουσίες για εκρηκτικές ύλε. Γι' αυτό θα εστιάσω την προσοχή μου σε αυτό. Αν δείτε το πακέτο στο σύνολό του, για μας τους πρασίνους έχει πολύ μεγάλη σημασία να δείξουμε ότι όταν καταπολεμούμε την τρομοκρατία θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και την επάρκεια των μεθόδων, έτσι ώστε να υπάρχουν αναλογικά μέτρα ε, με συγκεκριμένες εγγυήσεις για να μην υπάρχει παραβίαση των δικαιωμάτων των πολιτών. Με αυτές τις προτάσεις υπάρχουν ορισμένα θέματα. Αν δούμε πάλι το θέμα των πρόδρομων ουσιών, αν δείτε την υπάρχουσα νομοθεσία, την προϋπάρχουσα νομοθεσία, βλέπετε ότι δεν έχουμε αντιμετωπίσει το θέμα στο σύνολό του. Γι' αυτό χρειαζόμαστε περαιτέρω νομοθέτηση για να υπάρχει μια εξορρόπηση θεμάτων ασφαλείας και θεμελιωδών δικαιωμάτων. Όπως είπα και πριν, εμείς έχουμε ορίσει συγκεκριμένα, έχουμε ταυτοποιήσει προβλήματα. Δείτε το άρθρο 8, δείτε το προσεκτικά. Ήδη περνάει ο χρόνος και σε σχέση με τις ηλεκτρονικές αποδείξεις, τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία, είπατε ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν υπάρχει υποψία για έγκλημα. Μα πώς λειτουργεί αυτό έμπρακτα, τι χρειάζεται ε, δικαστική εντολή ή θα πρέπει να ζητήσει κανείς από τον Γενικό Εισαγγελέα ή το Δημόσιο Κατήγορο να ε, ζητήσει πληροφορίες. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω κατά πόσο ε, έχω κατανοήσει καλά το θέμα. Είμαι κάπως επικριτική με την ιδέα να μεταβεί κανείς ε, στις εταιρείες ή επιχειρήσεις απευθείας για αυτές τις πληροφορίες, γιατί θέτεται τον επιχειρηματία σε πολύ δύσκολη θέση θα πρέπει να δείτε πού υπάρχει η ρήξη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Σόφι Ιντβελτ και μετά η τελευταία ομιλήτρια, ο τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι δεν έχω τίποτα κατά της αρχής βελτίωση της δυνατότητας διενέργειας ερευνών. Αλλά η Ευρώπη αρχίζει από τη λάθος πλευρά. Δηλαδή, τώρα βγάζετε έναν κρίκο από την αλυσίδα και παράλληλα θέλετε να ενδυναμώσετε, να ενισχύσετε τα ε, δικαιώματα των πολιτών, προστασία δεδομένων, ιδιωτικότητα. Τι έχετε κάνει με την μηδενική εφαρμογή της ε, διαδικασίας αστυνόμευσης. Τι έχετε κάνει ως προς αυτή την ε, εφαρμογή. Σε ένα κράτος δικαίου Ίσως ε, χρειάζεται περισσότερος χρόνος, γι' αυτό υπάρχει και κράτος δικαίου και γι' αυτό υπάρχει προστασία των πολιτών. Είναι χρονοβόρα η διαδικασία. Και νομίζω ότι υπάρχει ένα θέμα με το κράτος δικαίου σε ορισμένες ε, χώρες. Τι θα γίνει με τις ε, αρχές της Ουγγαρίας, που πάει στη Γαλλία και λέει «Α, θέλουμε πληροφορίες για τον κύριο Σόρος» γιατί υποπτευόμαστε ότι έχει προβεί σε εγκληματικές ενέργειες. Τότε το Cloud Act είναι ο σύνδεσμος. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να κινηθούμε κατά τον ίδιο τρόπο με τους Ρώσους και τους Κινέζους όταν εγκρίνουν το Cloud Act. Και στις ε, συναναστροφές με τις ΙΠΑ έχω έχω χάσει κάθε εμπιστοσύνη στην ικανότητά σας να διαπραγματευτείτε. Δεν σας ενδιαφέρει παρά η φιλία σας με τις Αμερικανικές αρχές, όχι τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών και πολλές φορές αυτό ε, έχει να κάνει και με τις προσφυγές ενώπιον του ΔΕΚ και ευτυχώς είναι ο μόνος προμαχώνας προστασίας των δικαιωμάτων των ε, πολιτών. Είναι η μόνη αρχή που ίσως αποσοβεί στον κίνδυνο συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Αλλά εσείς δεν μπορείτε να κάνετε αναφορές σε συναλλαγές με τους Αμερικανούς. Δέχομαι την, το ζήτημα αρχής, αλλά θα πρέπει να απαντήσετε. Ε, για δύο λεπτά η τελευταία ομιλήτρια, η Άννα Γκόμες. Καλωσορίζω την αναθεώρηση αυτή γιατί δυστυχώς ε, ε, είχε ε, προϋπάρξει μια δύναμη πρόταση επιτροπής ε, την οποία είχαν αποστεώσει και τα κράτη-μέλη. Τώρα ε, λόγω Σάλισμπερι υπάρχει μεγαλύτερη όρεξη για δουλειά. Αλλά δυστυχώς ε, τα κράτη έχουν εγκλωβιστεί στα χρηματοπιστωτικά του συστήματα, δηλαδή με βάση ε, χρηματοπιστωτικούς κανόνες, ε, κανείς ε, στην ουσία δεν κάνει τίποτα άλλο από τα νόμιμοποιεί τους εγκληματίες. Θα κάνετε το ίδιο με αυτό που κάνατε για το PNR. Ποιες είναι οι υπόδομες. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλές φορές δεν έχουμε να κάνουμε ούτε καν με διοικητικά σώματα. Δηλαδή, τι κάνετε στην περίπτωση αυτή με τις ε, μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα για το πώς ε, θα αντιμετωπίσουμε τις FIU, δηλαδή τις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την πέμπτη οδηγία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τι θα γίνει ε, με τα κρυπτονομίσματα ή τα συγκεκριμένα παιχνίδια ε, τα επιγραμμικά παιχνίδια που δημιουργούν μεγάλη κερδοφορία. Μιλήσατε και για τις ταυτότητες. Τι θα γίνει όμως με τις χρυσές ε, βίζες, γιατί στην ουσία πουλάμε ε, διαβατήρια. Ο οποιοδήποτε κλεπτοκράτης θα μπορούσε να προωθήσει αυτά τα σχήματα και με τις χρυσές βίζες και με την νομιμοποίηση εσόδων. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για την συμβολή και το ενδιαφέρον σας σε αυτά τα θέματα. Ε, λυπάμαι για τη μορφή ε, της έκθεσης. Ε, βλέπω ότι υπάρχουν πολλές και διαφορετικές εισηγήσεις. Τρεις κανονισμοί, δύο οδηγίες, μία σύσταση σε, ένα, σε μία δέσμη μέτρων. Αναγνωρίζω ότι είναι πολλά. Αναγνωρίζω, όπως ε, είπε ο συνάδελφος, ότι θα πρέπει να εξηγήσουμε πώς ε, εντάσσονται αυτές οι προτάσεις σε μια γενική προσέγγιση. Πιστεύω ότι εντάσσονται εγώ. Είναι σχεδιασμένα είτε για να κλείσουν το χώρο στον οποίο ενεργούν οι τρομοκράτες ή μπορούν να ενεργήσουν οι τρομοκράτες και εγκληματίε, εγκληματίες ή να ε, ε, ενισχύσουμε την ανθεκτικότητά μας για να αντιμετωπίσουμε τις πιθανές επιπτώσεις αυτών των πράξεων και επιθέσεων και να ε, μπορεί να λογοδοτήσει κανείς. Είναι αυτό το πλαίσιο στο οποίο οργανώνουμε αυτά τα μέτρα και αυτά που έχω περιγράψει σήμερα νομίζω εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο. Είναι λεπτομερέστατα. Υπάρχουν αρκετά θέματα που προκύπτουν ε, και πρέπει να συζητηθούν επαρκώς. Δεν ε, θα μπορέσουμε να το κάνουμε εξαντλητικά. Ε, και απόψε και να καλύψουμε όλα τα θέματα, δεν νομίζω. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας ε, σε κάποια άλλη περίπτωση, είτε διμερός ή συλλογικός, όπως εσείς το θέλετε, να υψέλθουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Ε, σε θέματα συνομοθεσίας θα σίγουρα θα τα αναλύσουμε λεπτομερώς, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει πλήρη σαφήνεια. Ε, κάνω μια έκκληση σε εσά και με ενθαρρύνει η προσοχή που έχετε δώσει σε αυτά τα θέματα. Είναι να προσπαθήσουμε να ενεργήσουμε το ταχύτερο δυνατόν. Είτε θα πετύχουμε είτε όχι, αλλά θέλουμε να προσπαθήσουμε να δούμε, να περάσουμε από τα διάφορα στάδια αυτές τις προτάσεις μαζί, από κοινού σε αυτό το σώμα. Γι' αυτό ε, χαίρομαι που έχετε ήδη ορίσει εισηγητές και ελπίζουμε να υπάρχουν και οι και θα μπορέσουμε έτσι να προχωρήσουμε αυτό το έργο. Δεν είναι γιατί θέλουμε να προχωρήσουμε αργά ή να αποφύγουμε οποιαδήποτε θέματα, αντιθέτως. Τώρα, σε ένα ή δύο από τα σημεία τα οποία έχετε θίξει, δεν νομίζω να μπορέσουμε να καλύψουμε όλα τα σημεία που έχετε γύρει σήμερα. Και πάλι, χωρίς κάποια σειρά προτεραιότητας, στο θέμα των εκρηκτικών και των πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών. Προσπαθούμε να κάνουμε τους ελέγχους πιο πρακτικούς. Σε κάποιο βαθμό υπάρχει εναρμόνιση. Γιατί αρχικά, μέχρι σήμερα, Υπήρχαν τρία διαφορετικά πράγματα που μπορούσε να κάνει για, κανείς για να ελέγξει αυτές τις ουσίες. Είτε να τις απαγορεύσει, κάποια κρατημέλη το έχουν κάνει. Είτε να υπάρχει ένα σύστημα αδειοδότησης, άλλα κρατημέλη έχουν προπίσει αυτή την ενέργεια με κάποιους τρόπους εξάρτησης του σύστηματος αδειοδότησης ή με γραφές. Δηλαδή, ε, μέλη του κοινού μπορούν να υπογράψουν ε, και να αγοράσουν τις ουσίες ε, υπογράφοντας. Ε, εμείς πιστεύουμε αυτά τα μέτρα είναι πολύ χαλαρά για όλους τους λόγους που έχουμε προαναφέρει. Και από και στο εξή, τα συστήματα εγγραφή, όπω το τρέχον σύστημα στη Γαλλία, δεν πρέπει να εφαρμόζονται πια. Δηλαδή, είτε θα πρέπει να υπάρχει απαγόρευση, απαγόρευση αυτών των συγκεκριμένων ε, πρόδρομων ουσιών για τα μέλη του κοινού ή να υπάρχει ένα σύστημα αδειοδότησης και εκεί θα πρέπει να ε, θεσπίσουμε ένα πιο περιοριστικό σύστημα αδειοδότησης. Εδώ ε, το αντίβαρο εδώ θα πρέπει να είναι ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν διατάξεις για τους νόμιμους χρήστες αυτών των ουσιών, για σκοπούς εμπορικούς, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πρόδρομες ουσίες. Αυτά είναι τα προβλήματα τα οποία πρέπει να εξετάσουμε στη συνέχεια. Τώρα στο θέμα των δελτίων ταυτότητας. Και πάλι, προσπαθούμε να ε, λειτουργήσουμε αναλογικά. Αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα Μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση για τους αριθμούς, ε, αλλά οι μεγάλοι αριθμοί, ναι. Το πρόβλημα είναι ότι δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δελτία ταυτότητας, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν για να ταξιδεύουν, να εισέρχονται και να εξέρχονται της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν είναι βιομετρικά. Δηλαδή όλες οι προβλέψεις, οι διατάξεις τις οποίες συμφωνείτε για ελέγχους ε, στα εξωτερικά σύνορα, όλα αυτά τα μέτρα που συζητάμε για τον κώδικα του χορού Σέγγεν ε, και όλα τα μέτρα τα οποία επεξεργαζόμαστε μαζί δεν θα έχουν αποτέλεσμα για αυτούς που χρησιμοποιούν αυτά τα δελτία ταυτότητας που δεν είναι βιομετρικά. Άρα πρέπει να εξετάσουμε αυτό το πρόβλημα και να προσπαθήσουμε να βρούμε μια αναλογική λύση δεν θα εισηγηθούμε κάτι εδώ το οποίο δεν έχει ήδη συμφωνηθεί για την περίπτωση των διαβατηρίων. Άρα ελπίζω να βρούμε κάποιο τρόπο, μια ικανοποιητική λύση, αλλά υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να επιλύσουμε και πρέπει να δούμε πώς θα χειριστούμε ε, το θέμα των ανηλίκων. Υπάρχουν λεπτομερείς, ε, λεπτομερείς στοιχεία στην πρόταση. Αν θέλετε μπορούμε να τα εξετάσουμε λεπτομερέστατα μαζί. Στο θέμα της πρόσβασης ε, σε χρηματοοικονομικά στοιχεία και μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών FIUs. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάποιοι λένε ότι επειδή αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα με το, η τρομοκρατία χαμηλού κόστους, ε, ότι αυτό το, το οικονομικό μέρος είναι λιγότερο σημαντικό. Διαφωνώ με αυτό. Πρώτα απ' όλα υπάρχει μεγάλος αριθμός ε, χρηματοδότησης που είναι στα χέρια των τρομοκρατικών οργανισμών. Υπάρχουν ε, κονδύλια που χρηματοδοτούν τουλάχιστον στην κρίζα ζώνη ε, τους τρομοκράτες και θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε τα κονδύλια αυτά. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο δίκτυα FIU που να είναι τόσο ισχυρά. Θα πρέπει να τα ενισχύσουμε. Πρέπει επίσης να τακτοποιήσουμε σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση τους κανόνες σχετικά με την εμπλοκή των αρχών επιβολής του νόμου με τα FIUs και τις χρηματοπιστωτικές πληροφορίες διότι ε, κυμαίνονται από κάλεσε, όχι και τόσο καλέ. Θα πρέπει να ε, το κάνουμε αυτό ε, και ταυτόχρονα να είμαστε σαφείς και διαφανείς για τα θέματα προστασίας. Αυτός είναι ο στόχος μας ε, στις προτάσεις αυτές και προσβλέπουμε στην περαιτέρω συζήτηση μαζί σας. στη διαλειτουργικότητα τώρα, το οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε σε λίγο, πιστεύω, αλλά θα ήθελα να προκαταλάβω κάποια σημεία τα οποία έχουν ήδη εγερθεί. Εμείς εμπλέκουμε ε, την EDPS και τον Οργανισμό Θημεριωδών Δικαιωμάτων, τον ΦΡΑ, ε, σε θέματα διαλειτουργικότητα. Ε, είναι χάρη σε αυτούς τους οργανισμούς που έχουμε πετύχει θα εξετάσουν σε κάποιο μεταγενέστερο στάδιο. Έχετε δει τις εκθέσεις τους, ε, χρησιμοποιείτε τις εκθέσεις τους και εσείς θα πρέπει να εξετάσουμε στενά έτσι ώστε ε, να ε, δούμε ότι τηρούνται τηρούνται τα σχόλια από αυτούς τους οργανισμούς. Αλλά εάν είμαστε σε θέση μαζί να συμφωνήσουμε πάνω σε μία δέσμη μέτρων που να προβλέπουν ε, τις σωστές προστασίες, τότε ε, η υλοποίηση είναι το κλειδί. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα συνεχίσουμε από πλευράς Κομισιόν ε, να είμαστε αυστηροί σε θέματα υλοποίησης. Έχουμε τα τελευταία δύο χρόνια ενισχύσει την διαδικασία αναφοράς στο θέμα του συστήματος πληροφόρησης Schengen, για παράδειγμα, και κάποιες χώρες, όχι μόνο οι χώρες που αναφέρατε εσείς, αλλά κάποιες ορισμένες χώρες είχαν ε, σκληρές εκθέσεις για θέματα υλοποίησης του συστήματος Σέγγεν και ε, θα ζητήσουμε να λογοδοτήσουν όλες αυτές οι χώρες για να επανορθώσουν τα ελλείμματα που έχουν παρατηρηθεί. Αυτή, αυτό θα συνεχιστεί. Σημαίνει ότι θα πρέπει να επεκτείνουμε το στο πλαίσιο της διαλειτουργικότητας. Ε, δεν θα γίνεται απλά αναφορά στη χρήση ενός συστήματος ε, πληροφόρησης Schengen. Θα καλύπτει ε, όλες τις διατάξεις που έχουμε συμφωνήσει στα θέματα διαλειτουργικότητας. Στο θέμα των ηλεκτρονικών ε, αποδεικτικών στοιχείων. Υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία έχετε θίξει με τα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία πρέπει να συζητηθούν ε, λεπτομερώς και περαιτέρω, διότι είναι ε, σημαντική η δέσμη προτάσεων, αλλά ήθελα να πάμε ένα βήμα πίσω και να πούμε γιατί το κάνουμε αυτό. Γιατί όχι μόνο επειδή κάποιοι μηχανισμοί, φυστάμενοι μηχανισμοί, δεν ε, είναι τόσο κατάλληλοι όσο θα έπρεπε για την ε, φύση του εγκλήματος ε, στον κυβερνοχώρο και τις διερευνήσεις αυτών των εγκλημάτων, αλλά επίσης επειδή όποια και είναι η άποψή σας για τα MLATs, ε, υπάρχει Υπάρχει ο και περισσότερα αιτήματα για εθελούσια ε, συνεργασία. Γι' αυτό ούτε και οι δικαστικές αρχές, αλλά οι αρχές, η αστυνομία ε, ζητούν άμεση επαφή με παρόχο υπηρεσιών και ζητούν τη βοήθειά του. Μερικές φορές μπορεί να είναι αιτιολογημένο, αλλά είναι εκτός του πλαισίου των κανόνων και της διαφάνειας ο αριθμός ε, των ετοιμάτων για εθελούσια συνεργασία στο πλαίσιο των, ε, της αμοιβαίας δικαστικής ε, συνδρομής έχει πολλαπλασιαστεί επί 40 αυτή τη στιγμή. Πιστεύουμε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τις αρχές επιβολής του νόμου. Ε, στην συνέχιση των ερευνών τους, αλλά θα πρέπει να έχουμε ένα ε, σαφές ε, πλαίσιο με σαφείς κανόνες και σαφείς εγγύησεις στο θέμα της σχέσης με τις ΗΠΑ. Με απόλυτα σαφής ότι πρέπει να κάνουμε τη δικιά μας κατοικονεργασία. Θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι αυτό που κάνουμε εμείς λειτουργεί με βάση αυτά που έχουμε συμφωνήσει και ε, θα τα δούμε και ε, ως συνομοθέτες μαζί σας. Θα είναι μια ευκολότερη κατάσταση να έχουμε κάποιο διάλογο με τη ΣΥΠΑ αν έχουμε ε, σαφέστερη εικόνα της θέσης μας. Αν δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στο θέμα της δικής μας θέσης, ο κίνδυνος είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιδιώξουν να έχουν διμερείς σχέσεις με μονομενα κρατη κράτη-μέλη και θα επιδιώξουν να το κάνουν και αυτό θα προκαλέσει μία κατάσταση που δεν είναι ικανοποιητική. Στο τελευταίο συμβούλιο με το γεγονός ότι στη συζήτηση που ξεκίνησαν αυτοί, που δεν ξεκίνησαν με εμείς, τα ε, κράτη-μέλη υπογράμμισαν ότι ήταν σημαντικό να προχωρήσουμε με μια ευρωπαϊκή, ευρωενωσιακή θέση, γιατί αυτό ε, θα σημαίνει ότι είναι ξεκάθαρη η θέση μας και οποιασδήποτε εποφές γίνονται με τις ΣΥΠΑ θα γίνονται με βάση αυτής της συλλογικής θέσης Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είπανε τα κράτη-μέλη στο τελευταίο Συμβούλιο και απλά αναφέρω ε, τη συζήτηση που έγινε. Στο θέμα των άλλων ε, ζητημάτων που έχετε γύρει, δεν θέλω να ε, ξεπεράσω χρόνο μου. Μπορούμε ε, να κάνουμε κάποιες επαφές διμερώς για θέματα, για παράδειγμα, των χημικών, βιολογικών, ε, ραδιολογικών ε, απειλών και των μικρών και ελαφρών όπλων. Μπορούμε να το δούμε σε κάποια άλλη ευκαιρία όταν εκδοθεί η επόμενη έκθεση. Σοφή, με ακούς? Με μέτρο παρακαλώ. Ναι, όλες αυτές οι γενικές δηλώσεις περί της Θα ήθελα να ξέρω συγκεκριμένα, μετά από όλα αυτά που ακούμε για το GDPR, το δεύτερο τμήμα έχει ξεχαστεί εντελώς. Δύο κρατημέλη μόνο, μόνο το υλοποίησαν. Είναι τραγικό αυτό. Μας μιλάτε για αγγίσεις, ασφαλιστικές δικλείδες, μας λέτε ότι ζητάμε από τα κράτη-μέλη αν θα είχαν την ευγενή καλοσύνη να υλοποιήσουν. Όχι. Πρέπει να προσφύγετε την επομένη το πρωί στο δικαστήριο. Αυτό είναι μια έντονη αντίδραση. Ολοκληρώστε και θα συνεχίσουμε. Έχετε δίκιο που με πιέζετε όσον αφορά την εφαρμογή και την υλοποίηση. Αλλά Έχετε μάλλον λανθασμένες πληροφορίες όταν λέτε ότι δεν παίρνουμε στα σοβαρά την εφαρμογή και την υλοποίηση. Για το κάθε μέτρο, για όλα τα μέτρα και παραδείγματος χάρη για το θέμα των προσωπικών δεδομένων των επιβατών, το PNR, παρακολουθούμε εξαιρετικά προσεκτικά θέλουμε και για το GDPR να φτάσουμε στο επίπεδο που έχουμε φτάσει με το PNR. Αυτή είναι η πρόθεση της Επιτροπής. Κοιτάξτε, ναι, ε, χαίρομαι που ακούω αυτές τις πιεστικές ερωτήσεις, διότι πραγματικά έτσι πρέπει και με οδηγείτε να σας δώσω και τις απαντήσεις. Βεβαίως η ε, προσφυγή για τις παράβασεις θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και σαφώς και με ταχύτητα όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία θα περάσουμε στα επόμενα βήματα και δεν αστειευόμαστε με αυτό για κανένα από αυτά τα μέτρα. Δεν δέχομαι ότι για ένα συγκεκριμένο μέτρο ή σειρά μέτρων έχουμε διαφορετική ε, προσέγγιση από ό,τι για άλλες. Υπάρχουν οι εισηγητές για τα θέματα αυτά που θα συζητήσουμε τώρα που περιμένουν με μεγάλη υπομονή, οι σκιώδεις. Ευχαριστώ πολύ. Τους συναδέλφους πρέπει να περάσουμε αμέσως στην επόμενη συζήτηση το θέμα της διαλειτουργικότητας των συστημάτων και βεβαίως θα περάσουμε πρώτα με την νομοθετική διαδικασία. Έχουμε δύο εκθέσεις, Λένας και Πέλο. Θα ακολουθήσει ο Επίτροπος οι σκιώδες ζητώ συγγνώμη που περιμένατε και καθυστερήσαμε υπήρχαν όμως πάρα πολλές ερωτήσεις για το θέμα αυτό Θα σας δώσω λοιπόν το λόγο στους δύο σας και κατόπιν στον Επιτροπό. Ευχαριστώ. Εγώ πραγματικά δεν έχω τίποτα κανονίσει για σήμερα. Έχουμε λοιπόν χρόνο μέχρι να ολοκληρωθεί και η συζήτηση αυτή. Πρόκειται για τον εξυγχρονισμό του συστήματος πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βεβαίως έχουμε τα νέα συστήματα πληροφοριών, το ETS, το EQUIS και όλα αυτά που αφορούν και τις πληροφορίες που αφορούν τις θεωρήσεις. Οριζόντιο θέμα, όλα αυτά τα συστήματα πληροφοριών έχουν σχεδιαστεί σαν τελείως ξεχωριστά και διακριτά συστήματα. Βλέπετε εδώ παραδείγματος χάρη στο Στρασβούργο υπάρχουν οι περίφημοι σερβες το Eurodac, το σύστημα για τις θεωρήσεις, το ETIAS, το ES, όλα αυτά τα συστήματα είναι στον, στην ίδια αίθουσα, το ένα απέχει εκατοστά από το άλλο, δεν μπορούν όμως να επικοινωνήσουν. Δεν είναι συστήματα τα οποία μπορούν να ε, συνδυαστούν. Και πραγματικά επισκέφθηκα και στη Σικελία το σύστημα των hot spots που χρησιμοποιείται στα hot spots και στα σημεία εισόδου πραγματικά δεν είναι πλέον δυνατόν να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Η προτεραιότητα είναι πάρα πολύ σημαντική όσον αφορά την ασφάλεια. Είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Θα πρέπει λοιπόν επιτέλους να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που διαθέτουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα μέσα που διαθέτουμε, έτσι ώστε να γίνουμε αποτελεσματικοί περισσότερα στοιχεία αυτή τη στιγμή περισυλλέγουμε και δεν μπορούμε να τα συνδυάσουμε, να τα διασταυρώσουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε. Χωρίς λοιπόν να αλλάξει το σύστημα πρόσβασης και τα δικαιώματα πρόσβασης, καθώς και οι κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων, πώς μπορούμε να είμαστε πιο συστηματικοί, να έχουμε καλύτερη πρόσβαση στα συστήματα και αυτό για τους ειδικού, για αυτούς που εργάζονται στα σύνορα, που κάνουν τους ελέγχους, που πρέπει να διασταυρώσουν τα στοιχεία. Γιατί δεν μπορούμε να λαμβάνουμε σωστές αποφάσεις αν δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση. Με το συνάδελφο 191 τροπολογίες προετοιμάσαμε. 191. Μεγάλος αριθμός. Και εγώ ίδιος ξαφνιάστηκα. Πρόκειται για ένα τεχνικό θέμα, για ένα περίπλοκο θέμα και στηρίζουμε πραγματικά την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για όλα αυτά τα περίπλοκα θέματα. Υπάρχουν κάποια βέβαια σημεία που πρέπει να προσαρμοστούν. Το ένα είναι τα συστήματα αυτά πρέπει να εργάζονται ταυτόχρονα σε περίπτωση αν θέλετε προβλήματος του ενός και διακοπής ενός από αυτά τα συστήματα δεν μπορεί να μην υπάρχει backup, δεν μπορεί να μην υπάρχει η εγγύηση ότι το σύστημα θα συνεχίσει να λειτουργεί κάπου αλλού και είναι πολύ σημαντικό να μην υπάρχουν οι σημερινές αδυναμίες και ευαισθησίες του συστήματος. Επίσης, ο ρόλος και η δυνατότητα πρόσβασης της Europol. Ξέρετε ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να παραμείνει εκτός αυτού του συστήματος όλο το σύστημα πληροφοριών της Europol. Η Europol πρέπει να συνεχίσει να ολοκληρώνει τις αποστολές της, άρα ο διαλειτουργικός χαρακτήρας, η καλύτερη πρόσβαση των συστημάτων Europol και των υπολείπων είναι απαραίτητη. Τρίτον, οι προτάσεις που αφορούν αυτή τη διαλειτουργικότητα βασίζονται σε ελέγχους, βελτιώνουν τους ελέγχους, βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα. Την ίδια ώρα όμως οι προτάσεις αυτές μπορεί να επιβάλλουν επιπλέον υποχρεώσεις για αυτούς που διενεργούν τους ελέγχους στα σύνορα. Έχουμε λοιπόν υποβάλει προτάσεις για να υπάρχει ισορροπημένη προσέγγιση μεταξύ αποτελεσματικότητας και ε, συγκεκριμένης προστασίας και ασφάλειας. Τελευταίο σημείο, ο εντοπισμός συγκεκριμένων προσώπων, ο εντοπισμός κάποιων παραβάσεων. Είναι κάτι που σίγουρα θα πρέπει να γίνει με καλύτερη συνεργασία των κρατών μελών. μελών. χάρη υπάρχουν κρατημέλη που δεν μπορούν να μην ενισχύσουν, αν θέλετε, τους ελέγχους τον εντοπισμό των προσώπων στο σημείο εισόδου, πριν προχωρήσουν στις επόμενες διαδικασίες. Πιστεύω ότι όλοι οι συνάδελφοι γνωρίζουν απ' έξω τις 191 τροπολογίες και ότι τις επόμενες εβδομάδες θα μπορέσουμε να τις επεξεργαστούμε, να τις συζητήσουμε. Θα δώσω όμως αμέσως το λόγο και στο συνάδελφο, τον κύριο Μέλο. Κύριε Πίτροπε, θα μιλήσω πορτογαλικά. Βάλτε τα ακουστικά σας, παρακαλώ. Ε, Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους εκπροσώπους της που, με τους οποίους είχαμε εξαιρετική συνεργασία για να κατανοήσουμε θέματα ιδιαίτερα τεχνικά άρα δυσπρόσιτα και δυσερμήνευτα. Γιατί έπρεπε να κάνουμε μία προσπάθεια τεχνικής και όχι πολιτικής κατανόησης. Φαίνεται απόλυτα σαφές ότι θέλουμε να υπάρχει προστασία της ιδιωτικότητας. και δεν θέλουμε να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Και έτσι έχουμε καλύτερη ασφάλεια τηρώντας τις αρχές της ιδιωτικότητας. Και αυτή την προσπάθεια ε, έχει κάνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή για να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, να καταπολεμήσουμε την ε, τρομοκρατία, την παράνομη μετανάστευση και πολλά συναφή. Και πιστεύω ότι τα προϋπάρχοντα στοιχεία δεν θα πρέπει να ανταλλάσσονται για να αποφύγουμε τρομοκρατικές ενέργειες. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ανταλλαγή απόψεων και να μοιραζόμαστε αυτές τις ε, πληροφορίες για να αποσοβήσουμε κινδύνους. Και πιστεύω ότι δεν πρέπει να επαναλαμβάνεται η ιστορία στην αρνητική της έκφανση. Θα πρέπει λοιπόν να δεσμευτούμε όλοι έτσι ώστε να βελτιώσουμε αυτή την Ευρώπη όπου οι πολίτες θέλουν πρωτίστως ασφάλεια. Και γι' αυτό πιστεύω ότι τάχιστα θα πρέπει να διοχετεύουμε πληροφορίες στις αρχές ως προς τις μεταναστευτικές ροές, τις ενδυνάμει τρομοκρατικές ενέργειες και τις βάσεις δεδομένων όπου ε, καταγράφονται οι τρομοκράτες ε, με διαφορετικές ταυτότητες. Θα πρέπει λοιπόν να μπορούμε να ταυτοποιήσουμε τους ε, ενδυνάμει τρομοκράτες. Και γι' αυτό ανέκυψαν και τόσες ε, τροπολογίες λόγω ελήψεων. Και όλα αυτά τα είδαμε με τους ε, σκιώδεις για να υπάρχει συνεργασία μεταξύ Europol, ε, οργανισμού Διασφάλισης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και ούτω καθεξής. Και γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, Επιτροπή για τις ε, προσπάθειες που έχει καταβάλει και ελπίζω με τους σκιώδεις να φτάσουμε σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ και τους δύο εισηγητές για τη δουλειά. Όπως είπαμε, οι διερμηνείς δεν θα υπερβούν το ράριο τους. Θα κλείσουμε στις 10 ε, παρατέταρτο ακριβώς και λυπάμαι που καθυστερήσαμε στην έναρξη. Θα ζητήσω από τον Επίτροπο να μας δώσει τις πρώτες του αντιδράσεις. Είναι ένα πελώριο θέμα, αλλά αν θέλετε εν συντομία να αντιδράσετε σε αυτά που ακούσατε από τους ε, εισηγητές και από τους ε, σκιώδεις οι οποίοι θα ε, μιλήσουν εκ μέρους του κυρίου Νίτερ Μιούλερ και η Σοφή μπορεί να κάνει κάποια μικρή παρέμβαση. Επίτροπε παρακαλώ. Σύντομα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους, τους και τους σκιώδους. Ευχαριστώ για όλες αυτές τις ερωτήσεις. Ελπίζω αυτός ο διάλογος να είναι επικοδομητικός και καρποφόρος οι προτινόμενες ε, τροπολογίες ε, είναι προς μια πολύ χρήσιμη κατεύθυνση, είναι πικοδομητικές, θα πρέπει να ε, έχουμε να προστεύσουμε τα πράγματα, να, να βεβαιωθούμε ότι το σύστημα δουλεύει 24 ώρες, 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα, ότι υπάρχει backpack, ότι ενισχύουμε τα θεμελιωδή δικαιώματα χωρίς να απομακρυνόμαστε από τους στόχους που έχουμε θέσει. Ε, και ένα θέμα που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι πρέπει να πετύχουμε την κατάλληλη ε, πρόσβαση της, για την Europol. Αυτά είναι θέματα τα οποία σίγουρα θα τα προχωρήσουμε ε, καθώς διερχόμαστε τις 194 τροπολογίες. Θα ήθελα να αναφερθώ τις επικείμενες ε, προτάσεις ε, που θα προκύψουν είναι ένα σημαντικό θέμα. Κυρία Βίξτρομ, ήδη το έφυξε στην προηγούμενη συζήτηση. Ήδη επισημάνθηκαν στις προτάσεις του Δεκεμβρίου και θα παρουσιαστούν αυτή τη βδομάδα ε, στις 12 Ιούνιου, αύριο δηλαδή. Ή μάλλον την Τετάρτη θα παρουσιαστούν διορθώνει ο μιλητής έγιναν πολύ περιορισμένες αλλαγές για να ολοκληρωθεί η πρόταση του Δεκεμβρίου σε σχέση με το αίτια στο ΣΥΣ, το Ιουλίσα και για επικόστρου των χωρών σε σχέση με την διασύνδεση αυτών των συστημάτων με τις συνιστώσεις της διατηλουργικότητας. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει το Δεκέμβριο ε, γιατί οι διαπραγματεύσεις ε, δεν το επέτρεπαν σε εκείνο το στάδιο. Η Eurodac, ωστόσο, δεν έχει συμπεριληφθεί ε, στις τροπολογίες που θα προταθούν για να τις εξετάσετε την Τετάρτη. Και, όπως γνωρίζουμε, ε, η αρχιτεκτονική και του συστήματος Eurotac αυτή τη στιγμή δεν ε, μπορεί να ενταχθεί στο σύστημα διαλειτουργικότητας διότι αποθηκεύει μόνο βιομετρικά στοιχεία με ε, αριθμό αναφοράς αλλά κανένα άλλο δεδομένο προσωπικής ταυτότητας. Προτείναμε το 2016 ε, μια πρόταση για να το αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα, συμπεριλαμβάνοντας και στοιχεία ταυτότητας, αλλά επειδή κρεμεί ακόμη η συμφωνία σε αυτή την πρόταση της δεν ε, μπορούμε να προτείνουμε άλλες τροπολογίες για την Eurodac ε, σε σχέση με τη διαλειτουργικότητα αυτή τη στιγμή. Βεβαίω όλοι βλέπουμε τη σημασία ε, του να πετύχουμε ε, την ένταξη της Eurodac ε, στην αρχιτεκτονική της διαλειτουργικότητας. Και θέλουμε να συνεργαστούμε έτσι ώστε να το πετύχουμε το συντομότερο δυνατόν. Ελπίζω ότι ε, αλλιώς θα είναι, είμαστε σε θέση να δούμε αυτές τις ε, τροποποιητικές προτάσεις, θα να τις λάβουμε υπόψη ε, στα σχέδια των εκθέσεων που έχουν παρουσιαστεί. Αναγνωρίζω και εκτιμώ και συμμερίζομαι προσωπικά την επιθυμία ε, των εισηγητών και πιθανόν και ολόκληρη τη Επιτροπής ΛΥΠΕ να προχωρήσουμε με τακτικό τρόπο αλλά και ταχύ τρόπο ε, στις προτάσεις αυτές για να επιτευχθεί μια κοινή θέση πριν από το τέλος του μήνα με την επικείμενη Αυστριακή Προεδρία. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία για τριμερή διάλογο. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας μέχρι τις καλοκαιρινές διακοπές και θα είμαι στη διάθεσή σας και από τις αρχές Σεπτεμβρίου των Συντομών των Δυνατών. Μαζί μπορούμε να πετύχουμε τον κοινό στόχο να κλείσουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις μέχρι το τέλος του χρόνου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Προεδρία είναι εδώ. Να ξεκινήσουμε με τους σκιώδες. Κυρία Ντάλη, καταρχήν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Μπάλε και τον κύριο Λένα, του δύο συνεισηγητέ, οι οποίοι εργάστηκαν σκληρά για την έκθεση που μα υποβάλλεται σήμερα. Θα ήθελα παρόλα αυτά να μιλήσω για την έκθεση και τη δική μας στάση. Είναι σαφές για όλους μας αυτή τη στιγμή ότι όσο έχει αυτή τη στιγμή η πρόταση, κάτι που εμπεριέχει δεν μπορεί να προχωρήσει. Το δικαίωμα για ασφάλεια, το δικαίωμα για προστασία της ιδιωτικής ζωής μπορεί και πρέπει να συμβαδίζουν. Ακριβώς αυτό είναι ο σκοπός αυτής της νομοθεσίας να νιώσουν οι πολίτες ασφαλείς, αλλά η ασφάλεια σημαίνει ότι δεν θα μας παρακολουθούν, δεν θα μας εκτιμούν, ε, δεν θα μας κρίνουν σε σχέση με το χρώμα του δέρματός μας, τις πεπιθήσεις μας, τις ιδέες μας και σε κάθε περίπτωση κοιτώντας αυτήν την πρόταση βλέπουμε ότι θα γίνουν διαλειτουργικά τα συστήματα πληροφοριών στην Ευρώπη. Διαβάζοντας την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής της 17ης Απριλίου του 2018 ενσωματώνονται στοιχεία βιομετρικά, δακτυλικά αποτυπώματα για πάνω από 500 εκατομμύρια πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραβιάζονται εδώ το δικαίωμα, αν θέλετε, της ιδιωτικής ζωής και το τεκμήριο αθωότητας. Σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι προστατεύονται με το νομοθετικό αυτό κείμενο αυτές οι θεμελιώδεις ελευθερίας. Θα ήθελα να με πείσετε επίσης για το θέμα των 125 εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών που θα πρέπει να διασφαλιστούν με αυτόν τον τρόπο δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση ότι τηρείται η αναλογικότητα, η αρχή της αναλογικότητας μεταξύ του σκοπού που αποσκοπεί αυτό το νομοθετικό κείμενο και των μέσων που κινητοποιούνται. Σαφώς και οι αποφάσεις αυτές θα αλλάξουν εντελώς τον τρόπο ερμηνείας των ε, γνωμοδοτήσεων σε ένα σημείο το οποίο θα είναι για μένα αδύνατον να επιστρέψουμε στην προηγούμενη κατάσταση. Εννοείται ότι όλα αυτά τα συστήματα, η Europol, η Interpol, τα συστήματα που χρησιμοποιεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα που αφορούν την ταυτότητα, που αφορούν τα έγγραφα ταυτότητας, τα βιομετρικά στοιχεία τα οποία θα ενσωματωθούν, θα πρέπει να τα ξαναδούμε. Εκτός και εάν ενσωματωθούν ασφαλιστικές δικλείδες και εγγυήσεις εξαιρετικά σοβαρές και αυστηρές, διότι σε κάθε περίπτωση αν αποφασίσουμε να κάνουμε αυστηρότερους τους κανόνες θα πρέπει να τους κάνουμε και σαφέστερους. Αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να στηρίξουμε την πρόταση αυτή. Τέλος, τα νομοθετικά αυτά κείμενα απαιτούν μια εφαρμογή, μια τήρηση η οποία προϋποθέτει τον ενεργό και καθοριστικό ρόλο επιχειρήσεων και εταιριών πληροφορικής. Και σαν σκιώδης ηγητής χρειάζομαι πολύ περισσότερα σαφή και συγκεκριμένα στοιχεία που να αφορούν το ρόλο αυτών των επιχειρήσεων πληροφορικής. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Το λόγο θα δώσω τώρα στον σκιώδη της Γκουέ. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε επαναλάβει τους τελευταίους μήνες ότι χρειάζεται αυτός ο διαλειτουργικός χαρακτήρας. Ναι, το επαναλαμβάνουμε, το χρειαζόμαστε και πρέπει τα συστήματα να είναι συμβατά. Όμως, τι είναι πιο λογικό. Εγώ το εξετάζω αυτό όσον αφορά τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Βεβαίως χρειάζεται συμβατότητα συστημάτων και διαλειτουργικότητα. Εμείς σαν Ευρωπαίοι πολίτες τι ακριβώς χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε ένα συγκεκριμένο σύστημα, το ESP, παραδείγματο χάρη. Χρειάζεται ένα τέτοιο κανονισμό, δεν έχουμε πρόβλημα. Και δεν θα μιλήσω μόνο για διαλειτουργικό χαρακτήρα, από τη στιγμή που έχουμε αποφασίσει ότι το θέλουμε και το επιθυμούμε και μας εξυπηρετεί. Το CID, το MID, το CIR, όλα αυτά, αν τα κοιτάξω, διαπιστώνω ότι πρόκειται αποκλειστικά και μόνο για συστήματα τριτών χρονών. Το Eurodac, Βάσεις δεδομένων δηλαδή που αφορούν τα άτομα που έρχονται από τρίτες χώρες. Περί αυτού πρόκειται. Ρωτάω λοιπόν για ποιο λόγο, για ποιους λόγους θα να υπάρχουν σίγουρα καλή γνώμη προτείνεται κάτι τέτοιο. Ποια είναι τα στατιστικά δεδομένα τα οποία έχετε και σας οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Ποιες είναι οι βάσεις που διαθέτεται που αποδεικνύουν ότι οι απάτες όσον αφορά τα δελτία ταυτότητας και τα έγγραφα πιστοποιητικά είναι τόσο μεγάλες που να δικαιολογούν μια τέτοια πρόταση. Ένας, ένα σύστημα για να εντοπιστούν αυτοί που έχουν πολλαπλές ταυτότητας. Ένα άτομο δηλαδή το οποίο ενσωματώνεται με πολλές διαφορετικές ταυτότητες. Διασταύρωση στοιχείων λέγεται αυτό. Δεν μπορούμε να βρούμε ένα ουδέτερο σύστημα που να συνδυάζει τα υπάρχοντα. Γιατί εδώ βλέπω πολύ σοβαρές παρεμβάσεις στην ιδιωτική ζωή εκατομμυρίων πολιτών της Ευρώπης. Ακούσαμε από τους σοσιαλιστές την εκτίμησή τους. Εγώ σας λέω ότι είναι πολύ περισσότερα, πολύ περισσότερα άτομα των οποίων δεν προστατεύεται κανένα προσωπικό δεδομένο. Ακούσαμε εξάλλου κριτική και από ΜΚΟ οι οποίοι λένε με πολύ σοβαρό τρόπο ότι όλα αυτά δεν διασφαλίζουν απολύτως καμία προστασία των προσωπικών δεδομένων και τα εν, ενσωματώνεται όλα αυτά σε προτάσεις που αφορούν τη μετανάστευση. Πραγματικά δεν υπάρχουν ε, εγγύσεις, δεν υπάρχει η αναλογικότητα και την ίδια ώρα βλέπουμε ότι παραβιάζονται και οι εγγύσεις και τα προσωπικά δεδομένα και ήδη πιστεύω ότι χρειαζόμαστε πολύ περισσότερες επεξηγήσεις και εγγύησης. Ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος ομιλητής, η επόμενη ομιλήτρια. Η κυρία Βαλέρο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία και πιστεύω μάλλον θα ήθελα να έχουμε πολύ καλή συνεργασία ε, και στο μέλλον, αλλά τώρα θα πρέπει να τροποποιηθεί η πρότασή σας Έχουμε 194 τροπολογίες. Ελπίζω να μειώσουμε τον αριθμό αυτό δραστικά με συμβιβαστικές. Ένα από τα βασικά ζητήματα είναι το θέμα των διακρίσεων. Όπως είπα στις ε, προηγούμενες συζητήσεις, όταν μιλάμε για νέους κανόνες θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι ε, τα μέσα υπηρετούν τον τελικό σκοπό. Οι τροπολογίες μας σχετίζονται με εγγυήσει, αναλογικότητα και μέσα που υπηρετούν τον ε, απότερο στόχο. Υπάρχουν ε, και θέματα profiling, όπως είπε η Κορνέλια. Πρόκειται για ε, πολίτες τρίτων χωρών και όσους ε, φυσικά έχουν ζητήσει βίζα τύπου Σέγγεν και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να προσέχουμε θέματα διακρίσεων. Ένα άλλο θέμα είναι τι κάνουμε με τους Ευρωπαίους πολίτες που έχουν διπλή υπηκότητα. Ε, και κλείνω γιατί δεν έχουμε και πολύ καιρό. Ευχαριστώ. Ο Πίτερ Νίτερμιλ έχει το λόγο. Για τους σοσιαλιστές. Ο Πίτερ δυστυχώς δεν μπορεί να είναι εδώ. Και στα σχόλιά του θέλει να ευχαριστήσει όπως και η Μίρια τους δύο εισηγητές και αυτά που ουσιαστικά λέει είναι ότι είναι πάρα πολύ περίπλοκο το θέμα και αυτό το δείχνουν οι πολλές παρατηρήσεις που γίνονται. Είναι τεχνικό το θέμα, είναι περίπλοκο. Την ίδια ώρα όμως διαπιστώνουμε ότι άλλαξε η στάση μας σε σχέση με τη δημιουργία βάσεων δεδομένων που αφορούν την ασφάλεια. Η προηγούμενη προσέγγιση που ήταν ξεχωριστά συστήματα μη συμβατά μεταξύ τους μας οδήγησαν σήμερα σε μια κατάσταση από την οποία πρέπει οπωσδήποτε να απομακρυνθούμε για θέματα ασφάλειας και συνεργασίας. Αυτό που σήμερα όμως προτείνεται είναι να μπουν σε μία κοινή τράπεζα δεδομένων ενσωματώνοντας βιομετρικά στοιχεία κάτι το οποίο μας απομακρύνει πάρα πολύ από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ακριβώς επειδή το εύρος αυτής της αλλαγής είναι πάρα πολύ σημαντικό και επειδή υπάρχουν εκατοντάδες εκατομμύρια στοιχεία τα οποία αφορούν πολίτες τρίτων χωρών, θα πρέπει να δούμε καθοριστικό σημείο για μένα το θέμα της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θεωρούμε ότι δεν τηρείται η αρχή της αναλογικότητας με αυτή την πρόταση. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων των ε, σκιωδών εισηγητών ήταν σαφές ότι ένας από τους λόγους που ζητήσαμε να που μας ζήτησαν να συμφωνήσουμε με το να δημιουργηθούν ε, συστήματα με διαλειτουργικότητα και συνεργασία είναι για να παταχθεί το θέμα της απάτης σε θέματα ταυτότητας. Δεν έχω πιστεί ότι ένα πρόβλημα τέτοιο, του οποίου η, κλίματα, κλίμακα είναι πολύ περιορισμένη, δικαιολογεί την δαπάνη 500 εκατομμυρίων ευρώ για να παταχθεί. Θα ήθελα να υπενθυμίσω λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πολύ πρόσφατα μας έκανε μια σύσταση η Επιτροπή, δηλαδή να δημιουργήσουμε τρεις νέες τράπεζες δεδομένων, βάσεις δεδομένων. Ήδη λοιπόν συλλέγουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα με τον συνδυασμό αυτών των υπαρχουσών βάσεων δεδομένων απλώς θα δημιουργήσουμε μια τεράστια τέτοια βάση δεδομένων και αυτό που ζητάμε παραδείγματο χάρη είναι να επιλεγεί ο μακρύτερος χρόνος αποθήκευσης αυτών των στοιχείων από όλες τις προτάσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Χρειάζεται λοιπόν μια πολύ πιο προσεκτική και ισορροπημένη προσέγγιση. Μα ζητάτε να ακολουθήσουμε τελείως διαφορετικό δρόμο και για την πρόσβαση και για την υλοποίηση. Όσον αφορά το μητρό, το κοινό μητρό για την αποθήκευση των προσωπικών αυτών στοιχείων και τη δημιουργία μιας νέας βάσης δεδομένων, όσο και ε, να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε διαλειτουργικά συστήματα, θεωρούμε ότι αλλάζει πάρα πολύ σημαντικά η προσέγγιση μας. Ναι, έχουμε αργήσει, αλλά δεν φταίμε εμείς γι' αυτό. Δεν θα πρέπει να δεχτούμε και δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι αυτές οι αλλαγές προτείνονται είναι απλές τεχνικές λύσεις και προτάσεις. Πρόκειται για εξαιρετικά ευαίσθητα πολιτικά θέματα. Σύμφωνα με το άρθρο του 29 θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας έτσι ώστε όλες οι ανησυχίες που έχουν υποβληθεί να εξεταστούν προσεκτικά. Επαναλαμβάνω ότι όλα αυτά φαίνονται και στις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί. Θα συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε το θέμα αυτό με τους ε, συναδέλφους και οδησηγητές. Μια προσωπική παρατήρηση, κύριε Πρόεδρε. Όλα αυτά τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια, κατά κάποιο τρόπο με οδηγούν σε μια ερώτηση. Ποιο είναι αυτό το οικοδόμημα για την ασφάλεια που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε. Νιώθω κατά κάποιο τρόπο σαν το πουλί στο κλουβί. Δεν μπορεί να με φάει μια γάτα, αλλά τελικά δεν είμαι και ελεύθερο πουλί και αν κάποιος θέλει να τραγουδήσει και να εκφραστεί ελεύθερα δεν μπορεί και μάλιστα την ώρα που θέλουμε να σταματήσει να κελαϊδάει το πουλί του βάζουμε και μια κουβέρτα πάνω από το κλουβί του για να νομίζει ότι είναι νύχτα και να κοιμηθεί. Έτσι νιώθω. Οι διερμηνείς πρέπει να διακόψουν στις 21 ε, και 45 γιατί δεν θα γίνει καμία υπέρβαση. Η Σόφι Ιντβελτ. Πρώτο ερώτημα. Η Επιτροπή ή οποιαδήποτε γενική διεύθυνση συζήτησε το θέμα ε, διαλειτουργικότητας με μια εταιρεία που ονομάζεται Palantir. ή με άλλες εταιρείες και μπορείτε να μου απαντήσετε γραπτός. Θεωρείτε ότι αν συσταθεί ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να γίνει από μία εταιρεία ή εταιρείες που εντάσσονται στο ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο και όχι σε μία χώρα όπου θα υπόκειται σε ένα διαφορετικό καθεστώς κλητεύσεων. Και επίσης δεν σας κάνει εντύπωση ότι συνδέουμε όλες τις βάσεις δεδομένων μεταξύ τους αυτό είναι θετικό για την αστυνόμευση, αλλά νομίζω ότι η προστασία δεδομένων ε, είναι ένα θέμα εθνικής εμβέλειας. Μιλήσαμε για την οδηγία περί αστυνόμευσης. Εάν λοιπόν αν υποβάλλετε 10 τροποποιητικές προτάσεις γιατί η οδηγία περί αστυνόμευσης δεν μπορεί να εφαρμοστεί ή γιατί να κάνετε μία τροποποίηση και να περάσουμε σε έναν κανονισμό αφού δεν έχει, ε, δεν έχει σχίσει αυτό το σύστημα. Χολμάιερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ καταρχήν αυτό που βλέπω είναι ότι η πρόταση της Επιτροπής για την δημιουργία διαλειτουργικών συστημάτων είναι κάτι θετικό. Προστασία των δεδομένων. Προσπάθεια να δούμε αν με τη διασταύρωση των στοιχείων βελτιώνουμε το επίπεδο ζωής και την ασφάλεια των πολιτών μας. Αυτό είναι μια υποχρέωση που πρέπει να την ε, προσφέρουμε. Κάνω λοιπόν ανάποδα την ερώτηση στον Επίτροπο. Το θέμα του διαλειτουργικού χαρακτήρα των συστημάτων αυτών, όπως είπε και η συνάδελφος Σίπελ, βελτιώνει την αρχιτεκτονική των ε, συστημάτων αυτών. Θα πρέπει να στοχεύσουμε λίγο πιο πολύ τις προσπάθειές μας. Τα δεδομένα που έχουμε θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν καλύτερα, θα πρέπει να προχωρήσουμε στοχευμένα και να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα για να αυξηθεί η ασφάλεια των πολιτών μας. Να κάνουμε δηλαδή την βέλτιστη χρήση των στοιχείων που διαθέτουμε για προστασία των πολιτών. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, η διαλειτουργικότητα αυτή των συστημάτων Μπορείτε να μας πείτε πότε θα ολοκληρωθεί. Έχετε χρονοδιάγραμμα για τα διάφορα στάδια και το τελικό στάδιο ολοκλήρωσης. Για να μπορέσουμε και εμείς σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στηρίξουμε τη βελτίωση της αρχιτεκτονικής των συστημάτων πληροφορίας και με ισορροπημένο τρόπο ασφάλεια για τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και ισορροπημένη προσέγγιση. Οι διερμηνείς μπορούν να μεταφράσουν την τελευταία μου φράση. Λέει ο πρόεδρος. Σας παρακαλώ, σας εκλυπαρώ. Θέλω να πω στους δύο εισηγητέ, στους Κιώδης και στα υπόλοιπα μέλη. Ακούσαμε τις προτάσεις σας.